αλλά και βιώσιμη. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ψάρια στις θάλασσές μας, αν θέλουμε να είναι αποδοτική η αλία μας. Αυτό ισχύει και σε άλλους τομείς διατροφής για τη γεωργία, για καλλιεργειες Ισχύει παντού. Χρειάζεται ισορροπία δηλαδή στη φύση. Θα έλεγα μάλιστα ότι τα τρόφιμά μας στην Ευρώπη τα βρίσκουμε έτσι κι αλλιώς στη φύση. Για να έχουμε λοιπόν μια βιώσιμη αλία, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε έναν, μια ρύθμιση ελέγχων που θα σέβεται τις συμφωνίες στις οποίες έχουμε καταλήξει στο παρελθόν και μάλιστα συχνά μετά από μακρές νυχτερινές συζητήσεις. Πρέπει να σας πω ότι συχνά συζητάμε επί μακρό, καταλήγουμε σε συμφωνία μεταξύ φίλων, αλλά η συμφωνία αυτή στη συνέχεια πρέπει να τηρείται. Και αυτή είναι η μεγάλη μου προτεραιότητα για το φθινόπωρο, να καταλήξω σε έναν κανονισμό για ελέγχους που να δείχνει σε όλους και πάνω απ' όλα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι οι συμφωνίες τις οποίες έχουμε καταλήξει θα τηρούνται από όλους. Όταν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες του κανονισμού για τους ελέγχους, πρέπει να προσέχουμε πολύ την ε, αλία μικρής κλίμακας και την αρασιτεχνική αλία. Θέλω λοιπόν ο κανονισμός αυτός να είναι αποδοτικός, δηλαδή να ασχολείται και με την απόδοση της αλίας. Θέλω να αναπτυχθεί η αλία μικρής κλίμακας, γιατί είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Έχει κοινωνική αξία μεγάλη. Έχει μεγάλη σημασία για τον τουρισμό, για την παράδοση, γιατί την και τα έθιμα στις ακτές μας. Και άρα είναι αναγκαίο να την προστατέψουμε στο μέλλον. Δεν πρέπει δηλαδή να βάζουμε υπερβολικά πολλά βάρη σε αυτήν την αλία μικρής κλίμακας. Συνεπώς πρέπει να περιορίσουμε τη διαχείριση των ελέγχων έτσι ώστε να μην αποτελεί υπερβολικό φόρτο, υπερβολικό βάρος για την αλία αυτή. Οι πολίτες μας, από την άλλη μεριά, πρέπει να είναι πεπισμένοι ότι η Ευρώπη προστατεύει τη... τους ανθρώπους που ζουν στις ακτές και τους ανθρώπους που ζουν από την αλία. Όσον αφορά τώρα την υδατοκαλλιέργεια. Ναι, δεν αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου είναι αλήθεια. Όμως η Σουηδική Προεδρία δεν έχει βάλει, δεν είδε στην εμερήσια διάταξη κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά το θέμα αυτό. Αλλά ως αρμόδιος υπουργός πρέπει να πω ότι βλέπω μεγάλο δυναμισμό στον τομέα. Βλέπω να μπορεί να εξελιχθεί πολύ ο τομέας αυτός. Ό,τι γίνει όμως πρέπει να έχει σαν βάση την προστασία της βιοπικιλότητας των υδάτων μας και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας στον τομέα αυτό. Επίσης, μιλήσαμε για τις απορρίψεις νυχθείων. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, υπάρχει εδώ ένα συμβολικό ζήτημα. Είναι ακριβώς αυτό που δείχνει την αποτυχία της ε, κοινή ελευτικής πολιτικής. Για μένα πρόκειται για μεγάλη αποτυχία πράγματι, μεγάλη αποτυχία της πολιτικής αλίας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε ό,τι μέτρα χρειάζεται προκειμένου να μειωθεί αυτή η κατασπατάληση πόρων. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με τη μείωση των απορρίψεων. Κατά τις συζητήσεις μας πέρυσι με την Νορβηγία, συζητήσεις οι οποίες θα συνεχιστούν, ε, το θέσαμε αυτό το θέμα. Έπειτα με ρωτήσατε κάτι, να ε, δεν απατώμε, για την ολοκλήρωση κάποιων ε, συμφωνιών για προϊόντα που μας έρχονται από τις φώκες. Η τρέχουσα νομοθεσία προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις για την αλίευση φώκιας σε μικρή κλίμακα. Ελπίζω ότι θα λυθούν πάντως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ακόμα για τη Φιλανδία κυρίως, ίσως και για τη χώρα μου. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια όταν πρόκειται για την ελίευση φώκιας. Να την προστατεύσουμε δηλαδή περισσότερο. Τώρα, στη συνέχεια. πρέπει να δούμε το θέμα των αρμοδιοτήτων και πού είναι τα όρια μεταξύ των αρμοδιοτήτων των μεν και των δε. Καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα αυτό τίθεται όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει κάθε φορά που θέλουμε να θέσουμε κάποια όρια σε διάφορες χώρες και άρα πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, η τελευταία δυνατότητα θα ήταν στα πλαίσια της νέας κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ελπίζω όμως ότι θα βρούμε κάποια λύση νωρίτερα. Αλλιώ θα περιμένουμε τη νέα κοινή ελευθερική πολιτική. Για τις συμφωνίες μας με τρίτες χώρες τώρα. Ως Σουηδός Υπουργός Αλίας, Θεωρώ ότι χρειάζεται να καθορίσουμε αρχές για το μέλλον. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα εμπορικά ζητήματα, την εμπορική πτυχή και την ενίσχυση που δίνουμε με την περιφερειακή πολιτική. οι συμφωνίες που χρηματοδοτούνται από φόρους πρέπει να σταματήσουν. Ουσιαστικά, μάλλον για να το πω αλλιώς, όσον αφορά τις πιστώσεις ενίσχυσης, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν οι σωστοί έλεγχοι και θα λάβουμε υπόψη μας τους ελέγχους, τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Θα φροντίσουμε οι συμφωνίες αυτές να τίθενται σωστά σε εφαρμογή και να είναι αποδοτικές και για τις δύο πλευρές. Έρχομαι τώρα στον ε, κόκκινο τόνο. Εδώ το πράγμα, μάλλον τον τόνο, τον κοινό τόνο. Το πρόβλημα εδώ είναι μεγάλο. Υπάρχουν ε, ελλείψεις. Αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον, είναι η απόφαση να ληφθεί από όλες τις πλευρές. Θα έλεγα μάλιστα ότι υπάρχουν πολλά που χρειάζονται διευκρίνηση. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα σε επίπεδο συμβουλίου και έτσι να καταλήξουμε σε κάποια απόφαση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχουν ζητήσει άλλοι δύο συνάδελφοι το λόγο και μετά από αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τελείωσε ο χρόνος μας μαζί σας. Να δώσω καταρχάς λοιπόν το λόγο στον κύριο Στίβενσον, αντιπρόεδρο της Επιτροπής και ε, κατόπιν στον κύριο Κάντεκ. Κύριε Στίβενσον, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Προεδρεύοντα, ευχαριστούμε που είστε εδώ και για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ξέρω ότι είπατε ε, πως η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, επειδή θα πάρει χρόνο ίσως ε, δεν ε, πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικό θέμα της Προεδρίας σας. Ωστόσο, χτες ε, συζητήσαμε με τον Επίτροπο Μπόρκ, ο οποίος έχει, μας ανέφερε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για ένα τελείως καινούριο σύστημα διαχείρισης της αλίας. Δηλαδή, μας μίλησε για μεταβιβάσιμα δικαιώματα τα οποία δεν θα βασίζονται στα αλλιεύματα αλλά θα βασίζονται στην αλληλευτική προσπάθεια κτλ. κτλ. Θα τα ξέρετε φαντάζομαι όλα αυτά. Θα θέλαμε όμως από τη δική σας οπτική γωνία ή μάλλον από την ε, οπτική γωνία της Σουηδικής Προεδρίας να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα γιατί υποθέτω ότι θα γίνουν και διαβουλεύσεις και με τον τομέα για τα θέματα όλα αυτά. Ο κύριος Κάντεκ. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για τις απαντήσεις γιατί εν μέρη ουσιαστικά ε, μου απαντήσατε και εμένα στο ερώτημα που θα θέσω. Θα ήθελα θα θέλα εγώ, εκ μέρους και των άλλων Γάλλων συναδέλφων, να θέσω κάποιο ερώτημα στη Σουηδική Προεδρία. Επικεντρώσατε ή επικεντρώνετε τις προσπάθειές σας ε, στην Βαλτική θάλασσα ε, και αυτό το θέμα της Βαλτικής έχει συζητηθεί εκτενώς, αλλά υπάρχουν και άλλες θάλασσες και ο Ατλαντικός και, ο, ε, και η Μεσόγειος και τα λοιπά. Ε, και μιλήσαμε και για τα μικρά ψάρια εδώ και ακούσαμε τώρα, ακούσαμε και από τον Επίτροπο και από τον κύριο Στίβενσον εδώ να θέτει το θέμα των δικαιωμάτων αλίας που μπορούν να μεταβεβαστούν. Ε, αυτό είναι ένα θέμα ε, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες δυσκολίες ε, είτε οι μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις είτε τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα ε, μπορούν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σενάρια τρόμου για τους αλληλείς. Επίσης, εγώ όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα, στην ε, περιφερειακή προσέγγιση στην αλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η προσέγγιση, η διαφοροποιημένη αναπεριφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τη μικρή κλίμακος αλία και την υποστηρίζουμε. Δεν ξέρω αν η Σουηδική Προεδρία θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, ε, το θέμα των εισαγωγών σε σχέση με τα, την παραγωγή, αν θέλετε, των, ε, ε, τα αλλιεύματα των δικών μας αλλιέων, των Ευρωπαίων αλλιέων νομίζω ότι θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικές ακόμα απαντήσεις για το θέμα αυτό των εισαγωγών. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω και εγώ μια μικρή παρέμβαση κύριε Υπουργέ και κατόπιν θα σας δώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε. Εγώ, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλίας ως Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να σας πω ότι με χαροποιεί το γεγονός ε, ότι είπατε σήμερα ότι θα μελετήσετε επισταμένα τις προτάσεις ε, του Κοινοβουλίου μας. Ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε θέματα συναπόφασης, ε, τα οποία θα ζητηθούν ε, μεταξύ μόν και μόν και είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά και μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέσης οι οποίες λέγονται αυτή τη στιγμή ε, και το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να δώσει και τη σύμφωνη γνώμη του. Θα δώσει ένα ναι ή ένα όχι το οποίο θα είναι δεσμευτικό για το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως θα είδατε από κάποιες από τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν από τους συναδέλφους, ε, με τις συμφωνίες εταιρικής σύμπραξης. Μας ε, ενοχλεί λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών και έλλειψη διαφάνειας. Ε, κατανοούμε ότι για κάποια θέματα όπως είναι οι διαπραγματεύσεις, η αποκλειστική αρμοδιότητα είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούμε όμως μεγαλύτερη συμμετοχή και μία από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να είναι παρατηρητές στις μικτές επιτροπές για να δούμε λίγο πώς εκτελούνται, πώς διεξάγονται αυτές οι συμφωνίες αλίας. Και πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το αίτημα από πλευράς Κοινοβουλίου. Θα το ξαναδιατυπώσω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το Συμβούλιο είναι αυτό που δεν μας θέλει σε αυτές τις μικτές επιτροπές, αλλά πιστεύω ότι και από νομικής ε, σκοπιές ε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεν έχει καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να λάβετε υπόψη σοβαρά το αίτημά μας, διότι πραγματικά θα πολεμήσουμε προκειμένου να λάβουμε κάτι το οποίο θα ε, είναι το κατάλληλο και θα εξισορροπήσει λίγο αυτά τα πράγματα που αφορούν στην ενημέρωση και στη διαφάνεια και πολλοί βουλευτές θεωρούν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πληροφορίες, ότι γίνονται λάθος τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι λίγο, γίνονται λάθος τα πράγματα, υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ευαισθησίες, συγκεκριμένα πράγματα, αποχρώσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν να το λάβετε υπόψη, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Προεδρία Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε αγαστές σχέσεις. Εγώ ως Πρόεδρος ε, δεσμεύομαι γι' αυτό και σας εύχομαι ε, καλή επιτυχία και σας δω το λόγο για να απαντήσετε, διότι περατώθηκε νομίζω και η προθεσμία που είχαμε για σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. Tack för ordförande. Även i denna frågeomgång eh, tycker jag det är intressanta, viktiga och relevanta frågeställningar. Ναι. Ε, και σε αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων ετέθησαν πολύ σημαντικά θέματα και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να τα απαντήσω. Ε, μπορώ να πω ότι η Σουηδική Προεδρία θα ε, αναλάβει δεσμεύσεις και θα κάνει συζητήσεις εκτενείς για την και η αλληλευτική πολιτική και τα θέματα που αποσχολούν τον κλάδο της αλίας αλλά γιατί τελικά ε, χωρίς συζητήσεις και δια, διαβουλεύσεις δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε, ούτε καν σε κατευθύνες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πράγματι το εξάμεινο ή οι μήνες που απομένουν στην Σουηδική Προεδρία δεν μας δίνουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σημαντικά. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό ε, είναι να ορίσουμε κάποιες αρχές. Παραδείγματο χάρη, η αλία πρέπει να καταλήγει σε αλλιεύματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, και όχι σε παραλιεύματα. Εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να χρησιμοποιούμε τη θάλασσα, όχι να καταχρώμεθα των θαλασσίων υδάτων και της αλίας νομίζω ότι αυτές, αυτή η βασική αρχή μας βρίσκει όλους σύμφωνους προσωπικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ένα στοιχείο που σχετίζεται με την ε, μεταρρύθμιση βέβαια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, αυτό της περιφερειακής διαφοροποίησης νομίζω ότι πραγματικά αν δούμε αναπεριφέρεια τα θέματα και ε, θα τα αποκριθούμε σε ανάγκες περιφερειακές ε, ε, ειδικέ ε, τοπικές ανάγκες και αυτό είναι καλό. Τώρα το θέμα των δικαιωμάτων ελίε που μπορούν να μεταβιβαστούν και τα λοιπά, αυτό είναι μια τελείως καινούργια ιδέα που πρέπει να συζητηθεί ακόμη πολύ μικρή αλία, η μικρή κλίμακος αλία που αναφέρθηκε όντως είναι πρόβλημα και κοινωνικό και ενδεχομένως ηθικό πρόβλημα ε, αλλά και εδώ πρέπει να αναλύσουμε εκτενέστερα την κατάσταση πριν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νομοθετικές πράξεις. οι συμφωνίες τώρα εταιρικής σχέσης που αναφέρθηκαν και που περιλαμβάνουν ρήτρε εισαγωγή ε, προϊόντων από τρίτες χώρες κτλ. Σαν Σουηδός υπουργό Αλίας οφείλω να ομολογήσω ότι είναι σημαντικές οι συμφωνίες αυτές αλλά Νομίζω ότι απάντησα αυτό το ερώτημα ε, προηγουμένως, συγγνώμη. Ε, τώρα για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις μικτές επιτροπές ε, που έθεσε η Πρόεδρος ε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την συνθήκη της Λισαβόνας πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις για τις αρμοδιότητες, τη συναπόφαση κτλ. Εγώ ελπίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα περάσει και θα αρχίσει να εφαρμόζεται επί Σουηδικής Προεδρίας. Αυτό ελπίζω. Και τότε βεβαίως τα θέματα των αρμοδιοτήτων και εξουσιών θα διευκρινιστούν περαιτέρω. Ε, σας ευχαριστώ πάντως κύριε βουλευτές για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας, τα σημείωσα και πραγματικά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά κατά τον υπόλοιπο χρόνο της Σουηδικής Προεδρίας. En este momento, a ver, escúchenme, porque... Συγγνώμη, ακούστε με λίγο γιατί δεν με παρακολουθεί κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ κανένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας ενημερώσει για τα επόμενα θέματα. Ε, πέντε λεπτάκια λοιπόν ε, και συνεχίζουμε στις 10 και 10 για να κάνουμε τα υπόλοιπα θέματα. Σας παρακαλώ, οι λίγοι βουλευτές που είναι ακόμα παρόντες, ε, καθίστε για να ξεκινήσουμε με το σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Πριν όμως από το σημείο 12 θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ξανασυζητήσει το θέμα της ΝΕΑΦΚ, το οποίο χθε έμεινε σε κρεμότητα και θα συζητηθεί τελευταίο ε, στην ημερήσια διάταξη. Να ξεκινήσουμε όμως με το σημείο 12, πολιετέ σχέδιο για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού και για την αλληλεία του αποθέματος αυτού. Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Λίντεμαν, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κύριε Λίντεμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πρόταση της Κομισιόν από τον Απρίλιο του 2009 για το δυτικό απόθεμα Σαφρίδιου. Μιλάμε για βόρειο ανατολικό Ατλαντικό. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε λεπτομερή παρουσίαση. Θα σας κάνω μια παρουσίαση και θα σας μιλήσω και για τη σημασία αυτού του πολιωτού σχεδίου γενικότερα για την Αλία γιατί πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία για τις χώρες που α, αλλιεύουν στην περιοχή αυτή της θάλασσας. Ε, θα προσπαθήσω να δώσω και κάποια στοιχεία για το επιστημονικό υπόβαθρο της ε, πρότασης αυτής. θα σας περιγράψω επίσης και την εξέλιξη της πρότασης της Κομισιόν μέσω των διαβουλεύσεων με τον κλάδο. Έχει αρκετά κεφάλαια η πρότασή μας. Θα σας τα παρουσιάσω και τέλος θα σας πω και τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πώς συνδέεται αυτή τη στιγμή το πολιετές αυτό σχέδιο με τον κανονισμό τάκ και ποσοστώσεων γιατί αυτά τα δύο θέματα είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Να αρχίσω με τη σημασία νομίζω του σχεδίου αυτού για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Να τονίσω πρώτα πρώτα δύο πράγματα που για μένα έχουν μεγάλη πολιτική σημασία. Πρώτο, αυτό το πολιετές σχέδιο είναι πρωτοβουλία του τομέα, του κλάδου. Ε, είναι πρωτοβουλία του Πελαγικού Συμβουλίου εκεί, ε, από εκεί ξεκίνησε το πολιετές αυτό σχέδιο. Επίσης είναι καινοτόμο το σχέδιο αυτό όσον αφορά τους κανόνες αλίευσης που προβλέπει. Πώς εντάσσεται το πολιετές αυτό σχέδιο στην κοινή αλλιευτική πολιτική όπως ε, ξέρετε από την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ΔΟΘΕ η Κομισιόν εκπώνησε αρκετά πολυετή σχέδια στην αρχή επικεντρώθηκε στα αποθέματα τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και μετά ασχολήθηκε με αποθέματα τα οποία βρίσκονται σε λιγότερο κρίσιμη κατάσταση, αν μπορώ να το πω έτσι, και εδώ ανήκει και το δυτικό απόθεμα σε Το πρώτο σχέδιο που φτιάχτηκε για αυτά τα μη ε, κρίσιμα αποθέματα είναι το σχέδιο για τη Ρέγγα, δυτικά της Σκοτίας. Εγκρίθηκε φέτο το σχέδιο αυτό. Ήταν το πρώτο πολύετές σχέδιο για ένα πελαγικό απόθεμα. Και το πρώτο σχέδιο που σχετίζεται με πελαγικό απόθεμα σε ευρωπαϊκά ύδατα. γιατί τελικά τα πελαγικά είδη ε, είναι διασπαρμένα σε πάρα πολύ, πολλά ύδατα και η, άρα και σε ύδατα μη κοινοτικά. Ε, οπότε, ας πούμε για το σκόμβρο στην ε, στο βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό για τη Ρέγγα και τα Ήταν δύσκολο να οριοθετήσουμε τα αποθέματα στην, ε, στα κοινοτικά ύδατα. Μας περιπτώσει αυτό το σχέδιο της Ρέγγας ήταν το πρώτο για πλαγικό είδος στα ευρωπαϊκά ύδατα. Τώρα για το Σαφρίδι ε, και εδώ υπάρχει πρόβλημα οριοθέτησης αν θέλετε γιατί και η Νορβηγία ε, ενδιαφέρεται και για το είδος αυτό και έγιναν και πολλές συζητήσεις με την Νορβηγία για το πώς θα μπορούσαν τα πράγματα ε, να εξελιχθούν μακροπρόθεσμα, ποια θα ήταν η μακροπρόθεσμη αν θέλετε διαχείριση του αποθέματος αυτού δεν ε, Βεβαίως η Νορβηγία τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν αλλιεύει συστηματικά ε, το είδος αυτό ε, και τα αλλιεύματα τα νορβηγικά έφθυναν τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά ε, οι συζητήσεις με την Νορβηγία συνεχίζονται και με τις νήσους Φαρόε ε, και προβλέπεται, μάλλον συζητιούνται επίσης και ανταλλαγές ε, αλλιευμάτων με τις χώρες αυτές. Τώρα, γιατί προτείνεται εδώ πολύ σχέδιο του Σαφρίδη, γιατί προτάθηκε ένα τέτοιο σχέδιο γιατί πραγματικά είναι σημαντική σημαντικής, ε, μεγάλης οικονομικής σημασίας, ειδικά το δυτικό απόθεμα ε, σαφριδιού μεταξύ δηλαδή των πελαγικών ειδών που δεν γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση από κοινού με άλλες βόρειες κυρίως σκανδιναβικές χώρες ε, ε, το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού είναι το πιο σημαντικό από οικονομική άποψη άλλος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή η αλίευση του αποθέματος βρίσκεται κάτω από τα όρια του συνολικού επιτρεπόμενου αλλιεύματος, δηλαδή κάτω από το ΤΑΚ. Το απόθεμα βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση από άποψη υγείας αν θέλετε ε, είναι καλό και η συνέχιση αλίευση σε επίπεδο χαμηλότερο του ΤΑΚ νομίζουμε ότι θα, θα οδηγήσει σε πλήρη ανασύσταση του αποθέματος αυτού. Τώρα, ποιοι αλλιεύουν το σαφρίδι, ε, τα αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται είναι μεγάλα σκάφη από την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία πελαγικές τράτες επίσης από την Ιρλανδία ε, που έχουν ε, και δεξαμενές ψήξεις. Επίσης στην Ισπανία και στην Πορτογαλία υπάρχουν κάποιοι ε, που αλλιεύουν το απόθεμα αυτό, αλλά εδώ τα σκάφη είναι μικρότερα, οι επιχειρήσεις είναι μικρότερες και κυρίως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το σαφρίδι πουλιέται, εκφορτώνεται νοπό και που λέτε νοπό. Επίσης γίνονται εξαγωγές στην Αφρική και στην Ασία άσχετα από την ποιότητα του ψαριού. Άμα δούμε τώρα ποιες είναι οι αλληλευτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το απόθεμα αυτό. Οι για τις επιχειρήσεις αυτές το σαφρίδι είναι γύρω στο 10 με 20% του εισοδήματός τους, των εκφορτώσεων τους αν θέλετε. Όμως πρόκειται για ένα ψάρι το οποίο εκφορτώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή το 20% για το οποίο μιλάμε είναι σε απόλυτες τιμές μεγάλη ποσότητα. Βεβαίω οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται και με, αλλιεύουν και άλλα αποθέματα, παραδείγματο χάρη ε, ρέγκα, σαρδέλα, στα ισπανικά είδατε και άλλα απαλλαγικά είδη. Was die, ähm, Όσον αφορά τώρα τις ποσότητες εκφόρτωσης, ο μέσος όρος των τελευταίων ετών είναι 140.000 τόνοι, αρκετά μεγάλη ποσότητα δηλαδή. Τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην αλία αυτή έχουν ε, ποσοστώσεις δεδομένες η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τις μεγαλύτερες ποσοστώσεις και μετά ακολουθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Δυο λόγια τώρα για το επιστημονικά βιολογικά δεδομένα οι επιστήμονες ε, διαχωρίζουν τρία αποθέματα. Βόρειο, νότιο και δυτικό απόθεμα. Σαφριδιού. Το σχέδιο αυτό αφορά στο δυτικό απόθεμα που είναι και το μεγαλύτερο απόθεμα Σαφριδιού και το οποίο μελετάται ε, ιδιαίτερα από την Καταβρική θάλασσα μέχρι τα νορβηγικά ύλατα. Ήδατα εκτείνεται το απόθεμα αυτό, είναι πάρα πολύ εκτεταμένο δηλαδή, κυρίως στον Βυσκαϊκό κόρπο στην Καταβρική θάλασσα και στην ε, Βρετάνη ε, γίνεται η μεγάλη αλία. Πριν από μερικά χρόνια οι επιστήμονες ε, επαναπροσδιορίσαν την έκταση του αποθέματος αυτού γιατί υπήρχε ένα σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού που ε, ε, ε, προσπαθούσε να ορίσει ακριβώς τα αποθέματα σαυριδιού και έτσι στο τέλος της μελέτης αυτής οι ΆΙΣΕΣ και άλλοι οργανισμοί ε, επανα προσδιορίσαν το απόθεμα αυτό το οποίο ε, ε, μας ενδιαφέρει και το οποίο καλύπτεται από το σχέδιο αυτό. Το, από το 1982 και μετά ε, είδαμε στην περιοχή αυτή αύξηση σημαντική της βιομάζας και το 1983 βεβαίως υπήρχαν καινούργιες γενιές ε, μικρών ψαριών που έφτασαν στην περιοχή λόγω της αύξησης της βιομάζας βεβαίως εκείνη την ίδια χρόνια ε, οι αλλιεύσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και από τότε οι, οι ποσότητες που αλλιεύονταν κυμαίνονται σημαντικά από χρονιά σε χρονιά. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα οπόθεμα αυτό λόγω των κειμενωμένων ποσοτήτων που λιεύονται κάθε ε, χρόνο. Εκείνο που αποφασίστηκε είναι κάθε τρία χρόνια να γίνεται ένα survey που κυρίως γίνεται για το σκουμπρί αλλά θα περιλαμβάνει τώρα και το σαφρίδι για να συλλεχθούν περαιτέρω δεδομένα για τους επιστήμονες ούτως ώστε να προσπαθήσουμε μαθηματικά μοντέλα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αποθέματος. Ε, υπάρχουν κάποιοι βιολογικοί δείκτες για το απόθεμα αυτό ε, πριν από πολλά χρόνια με την Νορβηγία μαζί ανεπτύχθησαν οι δείκτες αυτοί. Βέβαια οι ISIS ε, μετά από το τελευταίο, τις τελευταίες μελέτες που έγιναν ε, είχε τις αμφιβολίες της για τους για τους δείκτες αυτούς το Πελαγικό Συμβούλιο το Πελαγικό ΡΑΚ ε, συνέστησε μια ομάδα εργασίας από από ειδικού για να ασχοληθούν και πάλι με τους δείκτες. Ε, ε, υπάρχουν πολλά μοντέλα για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς το απόθεμα. Τέλος πάντων έγινε μια πρόταση ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 μελετήθηκε και αξιολογήθηκε η πρόταση αυτή από τους δικούς μας τεχνικούς και από την ISIS ε, μας είπαν ότι το, η πρόταση αυτή μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί είναι συμβατή με τις βασικές αρχές οπότε ενθαρρυνθήκαμε κι εμείς και ως Κομισιόν και τελικά παρουσιάσαμε αυτό το πολιετές σχέδιο για το οποίο μιλούμε σήμερα. Για να δούμε πώς διαρθρώνεται το σχέδιο αυτό. Έχουμε το κεφάλαιο 1. Στο κεφάλαιο 1 αναφέρεται το, παρουσιάζεται το αντικείμενο του σχεδίου. Τονίζω ιδιαίτερα το άρθρο 2 που είναι το πεδίο εφαρμογή. Που ορίζει για ποιο σαβρίδι ακριβώς εφαρμόζεται το σχέδιο αυτό, δηλαδή ορίζει ακριβώς την έκταση του δυτικού αποθέματος. Ε, έχουμε ορίσει το δυτικό απόθεμα βάσει των επιστημονικών ε, στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ε, πρέπει να συμμορφώνονται η, συμμορφώνεται η έκταση που ορίζουμε εμείς εδώ με τα τάκ που ε, αποφασίζουμε κάθε χρόνο και εδώ δεν συμπίπτουν, θα επανέλθω σε αυτό στο τέλος της ομιλίας μου. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται το σχέδιο που μιλάει για πολιετή διαχείριση του δυτικού αποθέματος Αφριδιού. Μιλάει για υψηλές αποδόσεις Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν βιολογικά στοιχεία που να μας επιτρέψουν να είμαστε σαφείς για το πόση μπορεί να είναι η μέγιστη απόδοση ή το μέγιστο αλίευμα που μπορεί να αφαιρεθεί από το απόθυμα χωρίς να διακινδυνεύουμε ε, εξαφάνι, ε, εξαφάνιση ας πούμε του αποθέματος. Ε, το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει κάποιους κανόνες αλλιεύσης βάσει των οποίων ετησίως ε, υποπλογίζονται και τα στοιχεία και του Συμβουλίου. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρεται το θέμα των απορρίψεων Κοιτάξτε, εδώ ότι οι επιστήμονες μάλλον όταν έκαναν την πρότασή τους είπαν ότι μόνο αν καλύψουμε όλα τα αλλιεύματα σαφριδιού θα μπορέσουμε να, είμαστε, να έχουμε επιτυχία στην διαχείρισή μας για το απόθυμα αυτό. Οπότε εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη και απορρίψεις σαφριδιού. Ε, γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να γίνει μια εκτίμηση των απορρίψεων που εκτιμώνται γύρω στο 1 έως 5% περίπου και τελικά πήραμε μια μέση τιμή από τα τελευταία χρόνια εδώ. Ε, παρακάτω στα κεφάλαια 7, στο άρθρο 7 και 8 ε, αναφέρονται πιο περίπλοκοι κανόνες, στο 7 ιδιαίτερα αναφέρονται, αναφέρεται αναφέρεται τι πρέπει να υπολογιστεί για το survey, αυτό που πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια και η δυσκολία εδώ έγκυται στο γεγονός ότι ένα μέρος του ΤΑΚ θα πρέπει να είναι πρέπει να ορίσουμε ένα μέρος του ΤΑΚ που θα πρέπει ε, ούτως ώστε να είναι βιώσιμη η κατάσταση. Η ISIS ουσιαστικά όρισε μία μάξιμο ποσότητα της τάξης των 150.000 τόνων περίπου, δηλαδή το 50% του συνολικού, ε, των συνολικών τάξ ε, σαν βιώσιμο όριο και από εκεί και πέρα ε, το υπόλοιπο ΤΑΚ μπορεί να αλλιευθεί. Ε, εάν δούμε ότι το απόθεμα αυξάνεται, τότε μπορεί ε, να αυξηθεί και το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα προφανώς. Εάν δούμε ότι μειώνεται το απόθεμα τότε ε, το μισθό 50% του ΤΑΚ που δεν είναι βιώσιμο μπορεί έως και να μην μηδενιστεί. Υπάρχει και μια ανώτατη, ένα ανώτατο όριο, μια οροφή προς τα άνω πέραν του οποίου δεν ε, αυξάνεται υπερβολικά το κομμάτι του ΤΑΚ που μπορεί να αλληλευθεί. Τώρα, για τις χρονιές που δεν έχει γίνει survey των νοών. Ε, παρόλα αυτά ο, μπορεί κανείς ε, βάσει του άρθρου 6 να κάνει κάποιους υπολογισμούς για να προσδιορίσει ή να προσαρμόσει τα τάκ. Στο άρθρο 9 αναφέρεται ε, τι θα γίνει αν και εφόσον δεν υπάρχει μελέτη survey των όν παραδείγματος χάρη το τελευταίο έγινε το 2007 και σας λέω ότι αυτά τα survey γίνονται κυρίως για το σκουμπρί ε, αλλά παρεμπιπτόντως και για, από εδώ και μπρος θα γίνεται σίγουρα για το σαφρίδι τα παλιότερα στοιχεία δεν αναφέρονται όλα στο σαφρίδι. Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν χρειάζεται. Βεβαίως ε, εδώ μπαίνει και το θέμα του ιστορικού τάκ, το οποίο ε, ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν τάκ αναφοράς, διότι αν αναφέρεται στο στο ίδιο απόθεμα με την ίδια έκταση. Ναι. Αυτά τα ρυθμίζει το άρθρο 9 παράγραφος 2. Παρακάτω αναφέρονται κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται αν θέλουμε να αποφύγουμε ή να επιτρέψουμε αν θέλετε μια κατάσταση σαν και αυτή του 1982 ε, η 83 με την ε, με, μεγάλη αύξηση του γόνου ε, εκείνη την εποχή αύξηση βιομάζας αύξηση του γόνου κτλ και λέγεται πως θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τέτοια προσαρμογή για να ε, δούμε μήπως ε, πρέπει να αλλάξουν κάποιες βεσκές παράμετροι του όλου συστήματος. Ε, παρακάτω ε, αναφέρονται διατάξεις για τα σκάφη, τα λιευτικά τα οποία επιτρέπεται να λιεύσουν σαφρίδι, το άρθρο 12 αναφέρεται στους ελέγχους και στον κανονισμό ελέγχων. Αυτή τη, μιλάμε για το νέο κανονισμό ελέγχων όπου προβλέπεται έτσι και αλλιώ πως πρέπει να συγκρίνονται τα στοιχεία των διαφόρων κρατών μελών, διασταυρούμενοι έλεγχοι κτλ. Πολλαπλή έλεγχη. και τονίζεται ιδιαίτερα ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι για λανθασμένα δηλωμένες ποσότητες ή για λανθασμένο είδος που δηλώνεται, δηλαδή αντισκουμπρή σαφρίδι και τα ανάποδο. κατά πόσον τα σκάφη αυτά αλίευσαν στα ύδατα στο οποίο επιτρέπεται να αλίευουν γιατί τα μαλλιευτικά αυτά σκάφη μπορούν να λέγουν μόνο σε ορισμένα αποθέματα. Επίσης, στο, α, στο επόμενο άρθρο αναφέρεται ότι θα γίνει αξιολόγηση του όλου σχεδίου σε μεγάλο χρονικό διάστημα, 6 χρόνια αναφέρονται εδώ, αλλά εντωμεταξύ ε, θα γίνονται και τα surveys αυτά που σας ε, είπα ε, και θα παρακολουθείτε η κατάσταση. Στο άρθρο 14 τέλος αναφέρονται οι δυνατότητες ε, μέτρων στήριξης από το Ταμείο Αλίας όπου προβλέπονται δηλαδή οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης για μ, σχέδια πολυετή ανασύστασης, ε, δυνατότητες στήριξης λοιπόν και συγχρηματοδότηση από συγκεκριμένε συνθήκες και αναφέρονται συγκεκριμένα ε, στοιχεία αναφορά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να δούμε αν συντρέχουν οι περιστάσεις να δοθούν ε, ε για να δοθεί η συγχρηματοδότηση. Τώρα, να Είπα προηγούμενα ότι τον Απρίλη, ε, από τον Απρίλη, στον Απρίλη ανάγεται η πρόταση αυτή της Κομισιόν. Ε, και βεβαίως έχουμε συνέστηση του γεγονότος ότι η πρότασή μας αυτή απαιτεί την προσαρμογή των περιοχών ΤΑΚ και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα ε, στις ε, συζητήσεις και σε διαπραγματεύσεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Πρέπει να ε, υπολογιστούν και νέες ποσοστώσεις για τα διάφορα κράτη-μέλη και περιμένουμε βεβαίως ε, ε, και καινούργια επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα τα έχουμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο Βεβαίω ε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα είναι τα στοιχεία αυτά, δεν έχουμε και survey διάμεσα των αυγών των νοών. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πούν οι επιστήμονες τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ε, το σχέδιο αυτό βέβαια είναι τελείως καινούριο για τα κράτη-μέλη Ε, ξέρουμε ότι κάποια ξέρουν ήδη τα κράτη μέλη ότι ορισμένα κομμάτια της Κανταβρικής θάλασσας, ορισμένα κομμάτια της Βόρειας θάλασσας ή της Μάνχης θα πρέπει να ανακατανεμηθούν για τα ΤΑΚ. Ε, ελπίζουμε να βρούμε τη φόρμουλα που θα κάνει την προσαρμογή αυτή Ήδη έχει συζητηθεί εκτενώς το θέμα με τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι ε, το γεγονός ότι λέμε πως το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί από το 2010 και μετά, δηλαδή όταν θα εφαρμοστούν τα καινούργια τάξη και ποσοστώσεις, αυτό είναι καλό γιατί συμπίπτει η εφαρμογή αυτού του σχεδίου με τα καινούργια τάξη και κουότας και έτσι δεν υπάρχει αυτή η... Ε, δυσαναλογία αν θέλετε ή με αυτό το πρόβλημα όπου η έκταση του αποθέματος δεν συμπίπτει με την έκταση των τάξη. Ο Επίτροπος νομίζω αναφέρθηκε χτες στο γεγονός ότι ε, δεδομένου ότι θέλουμε όλα να εφαρμοστούν από το 2010 και μετά ε, αυτό σημαίνει πίεση χρόνου εμείς σαν ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να κάνουμε όση δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Ε, έχουμε ετοιμάσει σημειώματα για το πώς ε, εξελίσσονται ε, τα αποθέματα, τι στοιχεία έχουμε από τι τις μελέτες αυτές του γόνου και των νοών ελπίζουμε να βοηθήσουμε ούτως ώστε πράγματι να εφαρμοστούν όλα αυτά από το 2010 και μετά. Σας ευχαριστώ για την ε, λεπτομαρέστατη ε, παρουσίασή σας. Ο εισηγητής του θέματος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, αλλά θα το διαβιβάσουμε όλα όσα είπατε και θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να μιλήσει από αυτού. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Ε, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε επιτέλους μια πρόταση που συμφωνεί με τον ε, τομέα. Ε, δεν έγινε κάτι τέτοιο για την, με την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιετές πρόγραμμα για τον Μερλούκιο του Βορρά, όπου έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που είπαν οι περιφερειακές οργανώσεις Αλίας. Χαίρομαι λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε τη δέουσα ευαισθησία στο θέμα αυτό και μπορεί να προκύψει το θέμα αυτό ελπίζουμε να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εγκρίνουμε όπως το επιθυμεί και ο κλάδος αλλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και στη συνέχεια να περάσουμε στο σημείο 13 της ημερήσια διάταξης που είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο για το απόθεμα γάβρου στο Βυσκαϊκό κόλπο και για τι ελευθερικέ δραστηριότητε εκμετάλλευση του εν λόγω αποθέματο. Εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τον κύριο Πετιέρα από την Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να σας κάνω λοιπόν μία εισαγωγή για το μακροπρόθεσμο σχέδιο, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι βάσει αυτών που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές ε, είναι κατεπίγουσα η υιοθέτηση του θέματος ε, του σχεδίου αυτού πριν από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου διότι και ο κλάδος αλλά και το Συμβούλιο περιμένει τη συζήτηση ε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Συμβουλίου και να προχωρήσει ώστε την άνοιξη το καλοκαίρι του 2010 να έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει επίσης ένα ακόμα σημείο το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι τα καλά στοιχεία που μας έχει δώσει ο κλάδος. Ξεκινήσαμε με το σχέδιο αυτό εκ του μηδενός και ε, είχαμε πολύ καλά στοιχεία και από την γαλλική και από την ισπανική κυβέρνηση και συνεργαστήκαμε όλοι από κοινού μέχρι να υπάρξει μία συνένεση ε, για το τι θα πρέπει να επιλέξουμε για τους ε, κανόνες ε, ελέγχου, που είναι και αυτοί που θα σας παρουσιάσουμε εδώ. Μετά από αυτά λοιπόν, να περάσω στο περιεχόμενο της πρότασης. Να σας πω ότι η Αλία του Γαύρου από το 2005 βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της εξάλληψης του αλλιεύματος. Ε, το, ε, να σας πω εδώ ότι ο γάβρος είναι ένα ε, είδος το οποίο δεν ζει πολύ. Ε, είναι από αυτά τα είδη τα οποία επεκτείνονται πάρα πολύ αλλά και περιορίζονται πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου όταν βλέπουμε πότε έχουμε το ανώτατο και το κατώτατο σημείο. βρισκόμαστε λοιπόν στο ναδύρ εδώ πέρα του είδους. Και είναι πολύ καλό ε, να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ώστε να μην επιδεινώσουμε την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να καθορίσουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανταυτού που κάναμε μέχρι τούδες. Στις, ε, συνήθως στις συζητήσεις του Συμβουλίου λαμβανόντουσαν πολιτικές αποφάσεις και από εκεί και πέρα καθορίζονταν οι δυνατότητες για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία πρόταση η οποία θα βασίζεται στους ε, κανούς, ε, κανόνες ε, καλλιέργειας. Και θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια. Η στόχη του σχεδίου είναι καταρχής να διασφαλίσουμε ότι ε, θα έχουμε υψηλή απόδοση του γάβρου, ε, να έχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη σταθερότητα του πληθυσμού και να έχουμε χαμηλό κίνδυνο εξάλληψης του αποθέματος. θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από την αλία, να μπορέσουμε δηλαδή να αλλιεύουμε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να, ε, να διασφαλίσουμε ε, να είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα εξάντλησης του αποθέματος μέσα στην... Ε, στα επόμενα χρόνια. Έγινε μία μελέτη από μία ad hoc ομάδα από τη Γαλλία και την Ισπανία μελετήθηκαν ε, διαξοδικά οι διάφοροι κανόνες ε, καλλιέργειας και αυτό το οποίο λάβαμε με τη συνένεση και του κλάδου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το επισημάνουμε, είναι ότι οι κανόνες αλίευσης θα μπορούσαν ε, να εκφραστούν εδώ και με μαθηματικούς όρους, είναι πολύ δύσκολο βέβαια, απλά να σας το δώσω με λίγα λόγια. Ουσιαστικά το μέγιστο επιτρεπόμενο αλεύμα για το γάβρο, το οποίο θα ισχύει για τη χρονιά από την 1η Ιουλίου ε, της μίας χρονιάς μέχρι τις, την 30 Ιουνίου της επομένης, θα κλείνει μόνο εάν η βιομάζα ε, η οποία ελέγχεται την άνοιξη είναι λιγότερο των 40.000 τόνων. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ένα ελάχιστο επιτρεπόμενο αλίευμα, ένα ελάχιστο τάρκ των 40.000 τόνων. θα έχουμε ε, μία ακτίνα μεταξύ 24.000 μέχρι ε, και το BPA, το οποίο μετράται με κάποιον υπολογισμό και είναι το 30, ε, στις 33.000. Έχουμε και έναν παράγοντα εδώ, το γάμα που βλέπετε στην διαφάνεια, το οποίο πολλαπλασιάζει την τιμή της βιομάδας που έχουμε υπολογίσει αυτή την άνοιξη. Και σε αυτή την περίπτωση ε, το ποσοστό αλίευσης, το γάμα το οποίο προκύπτει εδώ, είναι στο 0,3, που σημαίνει ότι το 30% αυτού του αποθέματος της βιομάζας θα πρέπει να αλλιευθεί. Αυτό φυσικά θα φτάσει και σε ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα που θα είναι 33.000 τόνοι, που είναι το μέγιστο των εκφορτώσεων που έχουν καταγραφεί σε αυτή την ε, αλληλουχία μέχρι τούδε. The, Εφαρμόζοντας αυτό τον τύπο, έχουμε μία τιμή για το ποιο θα πρέπει να είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα στο παράρτημα 1 και μας δίνει και ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα ε, και για τη Γαλλία και για την Ισπανία. Αυτή η τιμή στη συνέχεια, όπως γνωρίζουν, γιατί ούτως ή άλλως βρίσκεται στον κανονισμό, αλλά κατόπιν θα διαβιβαστεί στα κράτη-μέλη και αυτή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί για κάθε κράτος μέλος για την ε, περίοδο αλίευσης του Γαύρου. Αυτό θα είναι το πρώτο κεφάλαιο του πολιετούς ε, σχεδίου. Το δεύτερο αφορά τους κανόνες ε, εποπτείας και παρακολούθησης οι οποίοι σαφώς θα πρέπει να συνάδουν με, τους με τον νέο κανονισμό εποπτείας τον οποίο συζητάτε και αυτό ε, θα καθορίσει και τι ακριβώς θα κάνουμε στα επόμενα κεφάλαια γιατί θα βασίζεται και στους βασικούς κανόνες, ε, κανονισμούς ελέγχου που θα έχουν υιοθετηθεί. Για να μην ε, περάσω σε κάθε άρθρο ξεχωριστά, να πω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια ειδική άδεια αλίας. Κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα, διότι ούτως ή άλλως η Ισπανία το έχει καθορίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Η Γαλλία όμως το χρειαζόταν ε, ε, νομίζω ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα έχουμε τα συστήματα παρακολούθησης σκαφών, τα VME, τα οποία θα πρέπει να έχουν ε, τεθεί σε εφαρμογή και αυτή είναι μια πολύ σημαντική ρήτρα. Μας λέει ότι το 1 τέταρτο του στόλου είναι κάτω των 15 μέτρων, που σημαίνει ότι δεν υποχρεωμένοι να έχουν σύστημα VMS. Εάν όμως αλλιεύουν γάβρο, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να καταγράφεται ε, το αλλιεύμα. Επίσης θα πρέπει να γίνονται διασταυρούμενοι έλεγχοι και όσον αφορά την αλλιευτική προσπάθεια και για, όσον αφορά το μέγεθος των αλλιευμάτων και γίνεται και ειδική μνήμα στην αλία με δόλωμα, η οποία δεν ε, προσμετράται μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία ε, από τον Ισπανικό στόλο για την αλία με δόλωμα που γίνεται ε, και στόχο κυρίως έχει το τόνο. Στο παράρτημα 2 και στο παράρτημα 3 έχουμε τα εθνικά προγράμματα δράσεων και ελέγχου τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν και τα οποία θα πρέπει να βασίζονται και στους κανονισμούς ελέγχων. Αυτά δεν είναι τίποτα καινούριο, είναι πράγματα τα οποία έχουμε ήδη σε εφαρμογή. Το τρίτο βασικό σημείο εδώ του προγράμματος διαχείρισης είναι η συνδρομή βάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάκτησης ε, βάσει και του κανονισμού 2371. Αν σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο εκτιμηθεί η βιομάζα και θεωρήσουμε ότι είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θα ισχύουν οι κανόνες για το πρόγραμμα ανάκτησης. Που σημαίνει προφανώς ότι έτσι καθορίζονται οι κανόνες για τις μέρες τις οποίες θα μπορούσαν ίσως να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας. Και τέλος, όποτε το επίπεδο της βιομάζας είναι πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ε, όριο, θεωρούμε ότι εκεί έχουμε ε, πρόγραμμα διαχείρισης και ακολουθούμε και τους ανάλογους κανόνες. Ένα από τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι όταν έχουμε πρόγραμμα ανάκτηση, έχουμε περισσότερε μέρε για χρηματοδότηση και έχουμε λιγότερε μέρε ε, εάν ε, εμπίπτουμε στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή έχουμε πρόγραμμα διαχείρισης, κάτι το οποίο είναι και λογικό. Στη συνέχεια του προγράμματος διαχείρισης, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, με τη βοήθεια και τη διαβούλευση των ε, περιφερειακών οργανώσεων ε, Αλίας, κυρίως των νοτιοδυτικών, ε, ΡΑΚ, θα μπορέσουμε να δούμε πώς αποδοτικό είναι το, πολυ... το μακροπρόθεσμο σχέδιο κάθε τρία χρόνια και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για κάθε ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ISIS σκέφτεται να κάνει μια συνεδρίαση benchmarking όπου θα αναθεωρεί τα σημεία αναφοράς και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάζει και την ανάλυση των κανόνων ελέγχου της αλίευσης, αλλά αυτό ε, θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Αυτά λοιπόν ε, ως ε, πρώτη εισαγωγή για το πρόγραμμα διαχείρισης. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η συγγήτρια, η κυρία Μπιλμπάου, θέλει το λόγο. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις εξηγήσει που μας δώσατε. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω εδώ λίγο, όπως φαίνεται και από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι τέσσερα χρόνια έχει κλείσει η Αλία, ότι οι ειδικοί εμπειρογνώμονε πίστευαν ότι πρόκειται για ένα είδος το οποίο θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε ως απόθεμα γρήγορα, σύντομα, χωρίς ε, ιδιαίτερο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό υπάρχουν επιπλέον παράγοντες όσον αφορά την αλία που μας οδηγούσε συμπεράσματα γιατί δεν αυξήθηκε το απόθεμα γάβρου. Οπότε, ίσως θα έπρεπε να αναλύσουμε σε βάθος με επιστημονικές μελέτες πού οφείλεται αυτό. Γιατί συμφωνώ στον κανονισμό με τον ορισμό ενός σχεδίου, συμφωνώ με τον έλεγχο, με την ρύθμιση, για το ότι πρέπει να είναι βιώσιμη αλία, που πρέπει να είναι και αποδοτική. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και καλά, αρκεί να έχουμε γάβρο να ψαρεύουμε. Ενώ αν δεν ξέρουμε γιατί δεν αναπαράγεται ο γάβρος όπως φανταζόμασταν νωρίτερα, ε, δεν θα ξέρουμε και ποιο θα είναι το μέλλον του είδους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε να δούμε τι άλλοι παράγοντες υπάρχουν που μας οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν έχει εξελιχθεί το είδος έτσι όπως οι επιστήμονες λέγανε ότι θα εξελίσσονταν πριν από πέντε χρόνια. Έπειτα τα τελευταία χρόνια αυτά ο κλάδος στο βυσκαϊκό κόλπο αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο κλάδος που αλλιεύει γάβρο είναι αλής μικρής κλίμακας. Ουσιαστικά γάβρο και τόνο. Και τέσσερα χρόνια τώρα δεν μπορούμε να ψαρέψουμε γάβρο. Επίσης, πίσω από τον κλάδο αυτό υπάρχουν ε, και πολλά άλλα χέρια εργασίας. Υπάρχουν ε, οι άλλες επιχειρήσεις, κονσέρβας για παράδειγμα, οι πάρα πολλές ε, γυναίκες που δουλεύουν στην αλία μικρής κλίμακας στον Βυσκαϊκό κόλπο Άρα καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί είναι μεγάλες. Διαπιστώνω ότι επαφές είχατε, αλλά δεν έχετε προσφέρει τίποτα στο κλάδο. Καλό θα ήταν στο μέλλον να έχετε άμεσε επαφές με τους ενδιαφερόμενους και το σχέδιο αυτό και οι εκθέσεις οι οποίες ετοιμάζονται να διέπονται από διαφάνεια. Ο κλάδος πρέπει να συμμετέχει ώστε οι επιστημονικές γνώσεις να μην είναι σε αντίφαση με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος στην πράξη. Οι επαφές αυτές είναι αναγκαίες, διότι αν προχωρήσουμε και θέλουμε ένα σχέδιο ισορροπημένο ανάμεσα στο τι μπορούμε να ψαρέψουμε και στην διατήρηση της βιομάσας, καταλαβαίνετε ότι σε λίγο δεν θα έχουμε κλάδο και δεν θα έχουμε τίποτα για να αλλιεύουμε. Αυτή η πρόταση κανονισμού είπατε ότι δεν έχει επιπτώσεις δημοσιονομικές. Μα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις οι δημοσιονομικές, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό για τους Δήμους στον Βυσκαϊκό κόλπο, πώς πλήττονται από την μη ανάπτυξη του κλάδου. Ποιες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κατάστασης αυτής τα τελευταία χρόνια, οπότε για το μέλλον να μπορεί να γίνει μια δημοσιονομική πρόταση. ώστε να μπορέσει ο κλάδος να διατηρηθεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές του στο μέλλον και να μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη αλληλεία μικρής κλίμακας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στίβενσον έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που μόλις ακούσαμε, πρέπει να δω όλη την κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε να ακούσουμε κάτι για τον κύκλο ζωής του Γαύρου. Δεν θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιοι άλλοι απειλούν τον ε, Γαύρο. Δηλαδή πέρα από την Αλία υπάρχουν άλλα ψάρια που επιτίθενται στο Γαύρο και καταστρέφουν τα αποθέματα. Όταν μας δείξατε τον μαθηματικό τύπο, ε, φάνηκε σαν να ήταν κάτι εύκολο να καταλάβει κανείς. Τώρα μπορεί μόνο εγώ να μην καταλαβαίνω. Έτσι αλλιώς ποτέ δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά στο σχολείο. Πάντως όταν είπατε ότι το BPA ήταν 33.000 τόνοι και αυτό είναι, το, είναι η προφύλαξη που έχουμε, τότε τα ανώτατα τάκ ποια είναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό καλά. Ίσως, όντως, εγώ να φταίω, αλλά δεν βλέπω Οπότε ίσως και το μαθηματικό τύπο να μπορέσετε να μας τον εξηγήσετε καλύτερα, με πιο απλά λόγια, για να καταλάβω εγώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, η κυρία Λέβιν έχει το λόγο. Uh, thank και εμείς με τα τεχνικά ζητήματα ασχολούμαστε, αλλά και με το θέμα τους κανόνες των ελέγχων. Αν πρόκειται και κάτω από 24.000, τότε είναι 0 τα τάκ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που είπατε. Πρώτον, όταν αναφερθήκατε στις δύο επιλογές για το σχέδιο διαχείρισης και το σχέδιο αποκατάστασης, ανασύστασης των ειδών. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τους τύπους. Μήπως θα μπορούσατε να μπείτε πιο πολύ στην ουσία. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τις δύο αυτές επιλογές. Εγώ δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Δεύτερον, Είναι δυνατόν ε, να συγκρίνουμε με κάτι αντίστοιχο για άλλα σημεία του κόσμου, για τον υπόλοιπο κόσμο, για το ίδιο θέμα πάντα βέβαια. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Ωραία, τότε και εγώ να κάνω ένα σχόλιο μετά από αυτά που είπατε. Η πρόταση αυτή, εγώ πιστεύω ότι προσπαθεί να λύσει το ζήτημα των ανώτατων ε, επιτρεπωμένων αλλιευμάτων όσον αφορά το γάβρο, να συμφωνήσει το Συμβούλιο κλπ. Λέτε ότι αυτό είναι ο στόχο τη πρόταση, αλλά συγχρόνω να εξασφαλιστούν τα αποθέματα του γάβρου. Πρώτα απ' όλα εξηγήσατε εσεί πολύ καλά ότι μιλάμε για πελαγιακό είδο που ζει τρία χρόνια και ότι έχει ένα... είναι κυκλική η περίοδο ζωή του. Όπω ξέρουμε, αυτό ισχύει στα πελαγιακά είδη. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε για την απόδοση που έχουμε για το είδος αυτό. Το λέω εξαιτία ε, αντικειμενικών δεδομένων. Αυτή είναι η βιολογία. Έτσι ζει το είδος. Ο γάβρος λοιπόν εξαρτάται από το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά. Και έχει φανεί, τουλάχιστον επιστημονικά, εγώ τέτοιες πληροφορίες έχω, ο ίδια δεν είμαι βιολόγος, ότι Εντάξει, δεν είναι μόνο για τον Μερλούκιο, αλλά με χαμηλή μάσα μπορεί να έχουμε καλή απόδοση. Η σχέση βιομάσα-απόδοση ε, για το Μερλούκιο δεν ισχύει, μάλλον που ισχύει για το Μερλούκιο δεν ισχύει και για τον Γαύρο. Αυτά είναι διατεραιότητες των ειδών. Αν λοιπόν με μια χαμηλή βιομάσα έχουμε καλή απόδοση και τότε καθορίσαμε τα μηδέν, τάκ, τότε η απόδοση αυτή, αφού σε τρία χρόνια θα πεθάνει ο γάβρος, τελείωσε. Δηλαδή, ο, η ζωή του γάβρου, όπως και άλλων πελογιακών ειδών, είναι πολύ διαφορετική. Φυσικά και χρειάζονται κανόνες για τα τάκ και σίγουρα εσείς προτείνετε καλύτερα πράγματα από αυτά που προτείνουν οι υπουργοί στο Συμβούλιο, που προτείνουν φρικτά πράγματα. Τα δικά σας μπορεί να είναι καλύτερα, αλλά αυτό το θέμα της απόδοσης δεν νομίζω ότι λέει πολλά πράγματα για το καθορισμό των ΤΑΚ. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για καλή διαχείριση του είδους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, αν μπορείτε να την απορρίψετε, να μου εξηγήσετε πώς. Λοιπόν, δεν έχει στήσει κανένας άλλος το λόγο, συνεπώς. Ο κύριος Φελτιέρα για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ε, ναι, ευχαριστώ. ξεκινήσω καταρχά από την παρέμβαση τη κυρίας Μπιλμπάου. Θα πρέπει να αναλύσουμε και τις αλλαγές στη βιομάζα, να κάνουμε κάποιες ε, μελέτες από αυτού. Πρόκειται για ένα θέμα ε, που αφορά στην επιστημονική μέθοδο. Ξέρουμε πολύ καλά τι μπορούμε να έχουμε με, την, ε, με το γάβρο στον Ειρηνικό ωκεανό στο Περού. Ε, όταν ε, έχουμε μεγάλους περιόδους στις οποίες εξαντλείται το απόθεμα του γάβρου ε, και περνάμε και μεγάλους, μεγάλες περιόδους στις οποίες έχουμε γάβρο για να χαρίζουμε κιόλας. Όταν όμως έχουμε ελνίνιο τότε εξαφανίζεται όλο το ε, απόθεμα γάβρου και επομένως ε, πρέπει να περιοριστεί και η αλληλεία του γάβρου στο Περού. Ε, γι' αυτό ακριβώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε πότε μπορούμε να αλλιεύσουμε και πότε όχι. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό που ακριβώς είπε η ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Προσπαθούμε να δούμε πιθανότητες. Ποια είναι η πιθανότητα να εκφαρμόσουμε ένα κανόνα ελέγχου ε, και η βιομάζα τον επόμενο χρόνο, αλλά και σε μία ακτίνα 10 ετών, να πέσει κάτω από το όριο που έχουμε θέσει εμείς ως ε, μέγιστη βιομάζα. Ουσιαστικά προσπαθούμε να το κάνουμε με συνεργασία αυτό, κυρίως για το γάβρο, ε, με, άλλα, με άλλες περιοχές η δυνατότητα να κάνουμε μελέτες, σαφώς υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες και φυσικά στο πρόγραμμα πλαίσιο θα έχουν ήδη γίνει κάποιες μελέτες, αλλά είναι προφανές ότι η αλληλεία, όπως είπε η κυρία Φράγα, εξαρτάται και από την ε, ε, από το απόθεμα και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, για παράδειγμα, αν είχαμε κλιματικές αλλαγές, ακόμα και μια μικρή αλλαγή θερμοκρασίας στην περιοχή στην οποία βρίσκεται ο γάβρος, ε, σαφώς θα έχει επιπτώσεις ε, στη θνησιμότητα των ε, ε μικρών γόνων ε, και φυσικά θα έχει ε, επιπτώσεις σε όλη την αλία. Εξακολουθούν να γίνονται διάφορες μελέτες και προσπαθούμε ε, να έχουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες ώστε όλα αυτά τα μοντέλα βάσει των οποίων συνεργαζόμαστε, τα πιθανοτικά μοντέλα, να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα και το πιθανό, η πιθανότητα σφάλματος να είναι μικρότερη. Τώρα, γι' αυτό που είπατε για τον κλάδο. Εγώ είχα μια πρώτη εμπειρία συνεργασίας με την ε, Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας του Νότου και ε, η συγκυρία ήταν εξαιρετική. Νομίζω και ο Ισπανικός και ο Γαλλικός ε, τομέας, κυρίως ο Βάσκικος τομέας που συμμετείχε στην, στην Περιφερειακή Οργάνωση, ήταν πάρα πολύ καλός και η συνεργασία ήταν τέλεια. Και η πρόταση, όπως είπε και η κυρία Φράγα, προέκυψε από τον κλάδο τον ίδιο. Οι πληροφορίες αυτές ε, περιγράφονται πάρα πολύ καλά και στην ανάλυση επιπτώσεων, η οποία λογικά είναι προσαρτημένη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για τον προϋπολογισμό, εγώ ειλικρινά βασίζομαι στην ε, ευρωπαϊκή βοήθεια, όπου, η οποία δόθηκε και στην Ισπανία και στη Γαλλία και φυσικά και στη βοήθεια που μπορούν να λάβουν από ευρωπαϊκής πλευράς ε, σε αυτά τα τέσσερα χρόνια που ε, θα έχουμε βιολογική πάυση. Τώρα, για τα όσα είπε ο κύριος Στίβενσον. Μου ζητήσατε να εξηγήσω λίγο πιο συγκεκριμένα τον κύκλο ζωή του γάβρου. Ο γάβρο, όπω σα είπα, είναι ένα είδο το οποίο ε, ζει πάρα πολύ λίγο, δεν ζει πάνω από 3-4 χρόνια και ε, ο κύκλος ζωής είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένος. Αναζητούνται κάποιες περιοχές ε, στις οποίες ε, το περιβάλλον είναι λιγότερο αλμυρό. Ο... Το μεγάλο ψάρι όταν πηγαίνει για αναπαραγωγή, πηγαίνει σε περιοχές στις οποίες έχει όσο το δυνατόν υψηλότερες ε, θερμοκρασίες. Ψάχνει περιοχές ε, στις οποίες θα είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία κοντά στην ακτή. Από το γόνο λοιπόν μέχρι το μεγάλο ψάρι έχουμε πολύ μεγάλη σχέση, συσχέτιση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αν έχουμε άνοιξη ε, και καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες για παράδειγμα, τότε έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή και το αντίστροφο. Ε, κάτι επίσης το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ είναι ο άνεμος. Σε περιοχές, σε περιόδους όπου έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, ε, Οπότε και έχουμε μεγάλη ανάμειξη των ε, υδάτων, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με την επιβίωση των ε, γάβρων. Και φυσικά όλα αυτά τα ε, πράγματα και η αναπαραγωγή για την επόμενη χρονιά μπορεί να επηρεαστεί. Και τελικά, όπως είπε και η κυρία Φραγκά, ε, ανάλογα με τις καιρικέ συνθήκες είναι τελείως διαφορετικό το τι θα έχουμε τη μία χρονιά σε σχέση με την επόμενη. Δηλαδή, ε, κυρίως έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τώρα, για τον κανόνα ελέγχου αλίευσης. Ζητώ συγγνώμη αν δεν ήταν ε, πολύ σαφής, ήταν λίγο απλοϊκή η εξήγηση που έδωσα για τον τύπο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι πολύ απλοί. Λέμε ότι αν έχουμε μία βιομάζα την οποία εκτιμούμε την άνοιξη ότι είναι κάτω από τις 40.000 τόνους, αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει να κλείσει η αλληλεία για αυτή τη χρονιά, αλλά όχι για τη χρονιά, για το έτος. Μιλάμε για περιόδους ε, για την ε, του γάβρου και μιλάμε από ε, για μια περίοδο από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου, γιατί σε εκείνο το διάστημα γεννιέται ο γάβρος. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν θα πρέπει να παρεμηνεύσουμε το BPA με το μέγιστο επιτρεπόμενο ε, αλίευμα. Άλλο είναι η βιομάζα που έχουμε στη θάλασσα και άλλο το μέγιστο επιτρεπόμενο ε, αλίευμα το οποίο αναφέρεται στο μέγιστο ποσοστό γάβρου που μπορούμε να αλιεύσουμε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός. Οι 33.000 τόνοι αντιπροσωπεύουν και το μέγιστο τάκ που μπορούμε να αλλιεύσουμε, αλλά και το BPA, το επίπεδο βιομάζας δηλαδή, στο οποίο θεωρούμε ότι ε, πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Πρόκειται όμως για δύο διαφορετικές έννοιες. Το ένα είναι η βιομάζα που έχουμε στη θάλασσα και το άλλο είναι αυτό που μπορούμε να αλλιεύσουμε. Νομίζω ότι ήταν σαφέ αυτό που είπε η κυρία Λεβάν για το Harvest Control Rule, για τον κανόνα ελέγχου της αλίευσης και για τις χρονικές διαφορές. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στο γεγονός ότι μέχρι τώρα είχαμε απόφαση για το μέγιστο επιτρεπόμενο ελίευμα το Δεκέμβριο για την επόμενη χρονιά ή ε, σε αυτό που θέλουμε να θέσουμε τώρα, διότι το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα καθορίζεται ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις που μπορούμε να έχουμε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και έχει να κάνει με τη βιομάζα που ε, εκτιμούμε ότι έχουμε την Άνοιξη. Να σας πω εδώ για όλα αυτά ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα όπου θα έχουμε μία ε, εκτίμηση το χειμώνα ή στο τέλος του χειμώνα για να δούμε λίγο καλύτερα τι γίνεται με την αναπαραγωγή, να μελετήσουμε λίγο καλύτερα, να δούμε αν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών, το επίπεδο βιομάζας από τη μία χρονιά στην άλλη. Δεν ξέρω αν αυτό απαντά σε κάποιο βαθμό σε αυτό που με ρωτήσατε. Τώρα, για τα άλλα μέρη του κόσμου, Αναφέρθηκα και στον, ε, γάβρο, στο μικρό γάβρο στην, ε, στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση και ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες, γιατί το φαινόμενο Ελνίνιο επηρεάζει όλες τις Αμερικανικές ακτές, και τις νότιες και τις βόρειες. Και το ίδιο θέμα έχουμε και στην, και στην Ευρώπη. Δηλαδή, το ίδιο φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στις ευρωπαϊκές αλλά και στις αφρικανικές ακτές. Ε, ε, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και στην Αμίμπια και στη Νότια Αφρική. Υπάρχει ένα είδος γάβρου που έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Και αυτό ακριβώς δυσχεραίνει την διαχείριση. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες ε, και διερωτώμαστε αν μπορούμε να έχουμε ε, συγκεκριμένους κανόνες για ένα είδος το οποίο είναι τόσο ποικιλόμορφο στη, ως προς τις ποσότητές του. Για να απαντήσω τέλος στην κυρία Φράγκα, ε, να πω ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τίποτα. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για πίνακες και για αναλύσεις κινδύνου, ουσιαστικά μιλάμε με πιθανότητες και φυσικά δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε τίποτα, αλλά τα επίπεδα των τάκ που καθορίζουμε, που προκύπτουν από τους κανόνες εκμετάλλευσης που καθορίζουμε εδώ, έχουν γίνει ή έχουν υπολογιστεί βάσει δεδομένων τα οποία συσσωρεύονται τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να εγγύθουμε τίποτα, αλλά Γι' αυτό ακριβώς και επιλέγουμε το επίπεδο εκμετάλλευσης. Αυτό το τελικό γάμα που έχει ο τύπος ε, έχει προκύψει βάσει μιας ανάλυσης κινδύνου. Βλέπουμε ποιος είναι ο κίνδυνος σε αυτό το πλαίσιο εκμετάλλευσης να πέσει το ποσοστό κάτω από την ε, ε, βιομάζα ή βλέπουμε μια πιθανότητα εξάντλησης, αν είναι πολύ ψηλή για παράδειγμα. Να πω εδώ ότι στην ανάλυση κινδύνου Εξετάζουμε μεν και το βιολογικό τομέα, αλλά στο περιθώριο έχει γίνει και μια οικονομική και κοινωνική μελέτη, τα, η οποία προκύπτει και στην ανάλυση επιπτώσεων. Ευχαριστώ πολύ για τις απεξηγήσεις ε, αυτές που μας δώσατε, κύριε Περτιέρα. Υποθέτω ότι η συγκίτρια με την γραμματεία θα φροντίσουν να καθορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες συνεδριάσεις μας και θα μας ενημερώσουν σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Και έτσι περνάμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης που είναι το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλλιευμάτων για τον τόνο. Είναι μια πρόταση που ετοίμασε η Επιτροπή με στόχο τις κοινοτικές προδιαγραφές βάσει απόφασης που έλαβε η ΚΑΤ ε, πέρυσι για καλύτερο έλεγχο των αλλιευμάτων του τόνου. Εφόσον συμφωνείτε κι εσείς, ο κύριος Κέμπ πρώτα θα μας εξηγήσει την πρόταση της Επιτροπής. Έχετε το λόγο λοιπόν και στη συνέχεια ο κύριος Ρωμέβα, ο εισηγητής, θα κάνει μια πρώτη παρουσίαση. Και μετά όποιος θέλει θα έχει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Oui, merci, Madame la Alors, comme vous l'avez Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε και εσείς, το πρόγραμμα αυτό τεκμηρίωσης θέλει να μεταφέρει στο κοινοτικό δίκαιο μία απόφαση της ΣΥΚΑΤ περσινή, σύσταση βασικά η οποία τροποποιεί προηγούμενη σύσταση που εγκρίθηκε το 2007, 07 2010 Αυτό το σχέδιο λοιπόν κανονισμού πέρα από την μεταφορά που είναι καθαρά νομικής φύσεως εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο καταπολέμησης ε, της ε, παράνομης και αδηλωτής αλίας. Η πρόταση ΚΑΤ λοιπόν απαγορεύει την αλία και τα, την παραγωγή προϊόντων που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις η ΚΑΤ. Το μέτρο αυτό που έχει εγκρίνει η ΚΑΤ αφορά βέβαια κύρια την αγορά. Έχει όμως επίσης ως στόχο να αντικαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βασιζόταν καθαρά στην εμπορία, δηλαδή στον έλεγχο των εισαγωγών και των εξαγωγών μόνο. Επρόκειτο για ένα σύστημα που βασιζόταν σε αυτό που ονομάσαμε τότε στατιστικό έγγραφο, που ενσωματώθηκε στο κοινοτικό δίκαιο, βάσει του 84-2003. Τώρα, όπως είπα και πριν, το σύστημα αυτό έλεγχε μόνο τις αγωγές και τις εξαγωγές. Δεν μας επέτρεπε να έχουμε άμεση σχέση με την ελίευση αυτή καθ' αυτή. Τώρα όμως, με το νέο αυτό πρόγραμμα, έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης των αλλιευμάτων με τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή το μερολόγιο πλοίου ή άλλα, αλλά και στην περίπτωση ειδικά του τόνου που είναι ένα είδος το οποίο παρευόμαστε πάρα πολύ διεθνώς, θα υπάρχει υπήρχε μάλλον το στατιστικό έγγραφο το οποίο παρακολουθούσε μόνο τις ε, διεθνείς συναλλαγές. Άρα είχαμε αλλιεύματα, εκφορτώσεις, εμπορία και από την άλλη μεριά ένα σύστημα παρακολούθησης των διεθνών συναλλαγών. Τώρα η φιλοδοξία του κειμένου και στόχος ε, του ΙΚΑΤ είναι τα δύο αυτά συστήματα να ενωθούν. Έχουμε ένα κοινό σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο να μας επιτρέπει να παρακολουθούν κάθε στάδιο της εμπορίας του τόνου από τη στιγμή της αλήψης μέχρι το τελικό στάδιο. Οπότε, ξέρετε ότι η αλία του τόνου είναι πολύ ειδική. Έχουμε και κλασικές πρακτικές, αλίευση, εκφόρτωση, πώληση σε ένα κράτος μέλος εκεί που έχουν εκφορτωθεί δηλαδή τα λιεύματα. Απ' την άλλη μεριά έχετε και δίκτυα εμπορίας πιο περίπλοκα, όπου εκεί έχετε την αλίευση ζωντανού τόνου, ο οποίος συνέχεια πηγαίνει σε κλουβιά για πάχυνση και μετά από αρκετούς μήνες πάχυνσης το προϊόν αυτό θανατώνεται και εξάγεται στην ασιατική αγορά, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία. Άρα λοιπόν έχουμε διαφορετικά συστήματα εμπορίας. Ο ε, Ικάτη, λοιπόν ήθελε να έχει μία και μόνη απάντηση. Ένα δηλαδή έγγραφο το οποίο να μας επιτρέπει, ένα έντυπο το οποίο να μας επιτρέπει να παρακολουθούμε ε, όλη αυτή τη διαδρομή. Θα σας εξηγήσω πώς έχει το σχέδιο κανονισμού. Λέμε καταρχήν ότι το πεδίο εφαρμογή, έτσι όπως παρουσιάστηκε του 94-2003 αναφέρεται στον τελωνιακό κώδικα για τον ε, τόνο τούνους τίνους. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα έγγραφα που αποτελούν και τη βάση του εγγράφου, επισυνάπτονται στο σχέδιο κανονισμού και είναι τα ίδια που έχουμε και στην απόφαση κάτι. Τα έγγραφα αυτά λοιπόν αποτελούνται πρώτον από το έγγραφο αλίευσης του τόνου. Αν δείτε το έγγραφο στο παράρτημα 3 του σχεδίου κανονισμού μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε όλα τα σχέδια όπως είπα και πριν από την αλίευση, την εμπορία, τη μεταφορά του τόνου όταν πρόκειται για ζωντανό τόνο, τη μεταφορά λοιπόν, την καλλιέργεια, σας είπα πριν ότι έχουμε και πάχυνση την ε, σφαγή και στη συνέχεια τα εμπορικά δεδομένα, δηλαδή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ε, παρουσία στην προέλευση του προϊόντος και πού απευθύνεται, ο προορισμός του. Αυτό λοιπόν το ενίο έγγραφο αποτελεί και τη βάση του συστήματος. Σε επίπεδο ΙΚΑΤ πρόκειται για πρόγραμμα αλίευσης, καταρχήν αυτή είναι η βάση και όπως θα δείτε και στο σχέδιο κανονισμού, υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Γιατί άλλος ασχολείται με την ε, αλίευση που είναι ο πλοίαρχος, έτσι ο καπετάνιος του σκάφους που κάνει την αλίευση, αλλά μετά υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι όταν πρόκειται για την πάχυνση, για την εξαγωγή. Και εδώ η επεύθυνη της ηχθειοκαλλιέργειας ή της εξαγωγής αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Όσον αφορά την συμπλήρωση του εγγράφου, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πρέπει να γράψουν στο έγγραφο την προέλευση του προϊόντος, το όνομα του σκάφους δηλαδή, και όλες τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την προέλευση του προϊόντος, αλλά και τον προορισμό του. Για κάθε τμήμα που συμπληρώνει ο καθαρμόδιος, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στο σύστημα, ε, πρέπει να υπάρχει και επικύρωση για την κάθε πλευρά από τις εθνικές αρχές. Το ελέγχουν αυτό δηλαδή οι εθνικές αρχές. Η βασική αρχή εδώ είναι ότι ο κάθε αρμόδιος είναι υπεύθυνο για τη συμπλήρωση των γράφων. Χωρίς να πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, ε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες υποχρέωσεις και κάποιες απαγορεύσεις. Από τη στιγμή όπου ζητάτε την επικύρωση ενός τέτοιου εγγράφου, αναλαμβάνετε τη δέσμευση κατά κάποιο τρόπο, να μην βάζετε τόνο εκεί που δεν πρέπει και να μην προμηθεύεστε από σκάφη τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ΙΚΑΤ. Τα κράτη-μέλη από την άλλη μεριά που είναι υπεύθυνα για τα έγγραφα αυτά τελικά, αναλαμβάνουν την ευθύνη να μας δίνουν τα έγγραφα από σκάφη τα οποία έχουν αδειοδότηση. Για την επικύρωση γίνεται από τις εθνικές αρχές που καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Οι επικυρώσεις αυτές λοιπόν γίνονται με υπογραφή, σφραγίδα, επίσης και επίσης η επικύρωση αυτή άρρητα σημαίνει ότι οι αρχές επαληθεύουν ότι είναι αδειοδοτημένο το σκάφος για τη συγκεκριμένη αλία, ότι οι ποσότητες που ολιεύθηκαν όντως είναι σύμφωνες με τις ποσοστώσεις κλπ. κλπ. Επίσης, ο κατάλογος, ο κανονισμός κατάλογος αναλαμβάνει διάφορες αρχές που πρέπει να τηρούνται πριν βάλει ο υπεύθυνο στην υπογραφή του για επικύρωση στο έγγραφο. Τώρα, ε, μια μικρή εξαίρεση, τα κράτη-μέλη. Μπορούν, αν θέλουν, να μαρκάρουν το κάθε ψάρι. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένες χώρες που θέλουν να έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Αυτές δεν χρειάζεται να δίνουν επικύρωση. Δηλαδή το έγγραφο γενικά χρειάζεται επικύρωση, αλλά όταν ο αλίεας βάζει σφραγίδα στο ψάρι, τότε δεν χρειάζεται επικύρωση. Αυτή είναι μια μικρή εξαίρεση στην επικύρωση. Κατά τα άλλα, το σύστημα παραμένει ίδιο. Έρχομαι τώρα στο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την επανεξαγωγή. Εδώ εξετάσαμε το δεύτερο έγγραφο, που είναι το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλευμάτων για τον τόνο. Ε, έχουμε την περίπτωση λοιπόν της επανεξαγωγής, οπότε προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, προϊόντα που έχουν αλλιεύσει σκάφη Λιβύης ή Τινησής και που έχουν μπει σε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται για εισαγωγή, έτσι. Είναι ένα παράδειγμα που σας δίνω. Από τη στιγμή λοιπόν που τα προϊόντα αυτά πάνε για καλλιέργεια, πάχυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξαχθούν μετά στην ασιατική αγορά, τότε το έγγραφο αλίευσης πρέπει να συνοδεύεται από ένα δεύτερο έγγραφο που είναι το πιστοποιητικό επανεξαγωγής. Με αυτά τα δύο έγγραφα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε. Όχι μόνο την προέλευση του προϊόντος που εισάγεται, αλλά επιπλέον έτσι μπορείτε να ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι ποσότητες που επανεξήχθησαν στη συνέχεια. Επίσης, μπορεί να εξάγεται μία μικρή ποσότητα της αρχικής που έχετε εισαγάγει. Χάρη λοιπόν σε αυτά τα δύο έγγραφα γνωρίζετε με ακρίβεια τι έχει επανεξαχθεί και τι παραμένει στην καλλιέργεια πάχυνσης. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν εισάγεται ας πούμε 100 τόνους ζωντανού τόνου, δεν εξάγεται απαραίτητα 100 τόνους, γιατί είναι η πρακτική εμπορίας τέτοια που οι ποσότητες κερματίζονται και δεν φεύγουν ολόκληρες. Το έγγραφο αυτό είπαμε πρέπει να επικυρώνεται σύμφωνα με τους ίδιους τρόπους όπως και το έγγραφο αλίευσης. Στο κεφάλαιο 4 είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πέρα από τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν το εμπόρευμα, είναι ζωτική σημασία όχι μόνο τα κράτη-μέλη μεταξύ του, αλλά και τα κράτη-μέλη με τα άλλα συμβαλόμενα μέρη, γιατί πρόκειται για μια αγορά, όπω σα είπα, όπου συμμετέχουν ε, πολλοί παράγοντες και από τρίτες χώρες. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει μεταξύ τους να επικοινωνούν και να μπορούν να κάνουν επαληθεύσεις. Άρα λοιπόν ε, μεταφέρεται και το έγγραφο και ανακοινώνεται, αλλά επίσης κάθε φορά που χρειάζεται μια επαλήθευση. Αν δηλαδή ένα κράτος μέλος έχει μια αμφιβολία για την επικύρωση ενός εγγράφου ή για την νομιμότητα κάποιων αλλιευμάτων, πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους για να αρθεί όποια αμφιβολία υπάρχει. Αλλιώς μπορεί να μπλοκαριστεί η συνέχεια της διαδικασίας, η μεταφορά ας πούμε του τόνου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται παληθεύσεις για να επιβεβαιώνονται ή όχι οι αμφιβολίες. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό των επαληθεύσεων. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σημεία επαφής, τα οποία αναφέρονται στο, στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΤ. Το κεφάλαιο 5 αναφέρει, είπαμε, τα σημεία επαφής τις λεπτομέρειες των αρχών που πρέπει να επικυρώσουν τα έγγραφα. Όταν, και εδώ συγκεκριμένα, ένα κράτος μέλος, ένα ευαλόμενο μέρος, ορίζει κάποια αρχή αρμόδια για την επικύρωση των εγγράφων, τότε η πραγματοποίηση της επικύρωσης αυτής, δηλαδή το όνομα, υπογραφή, η σφραγίδα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή κάτι. Άρα, άπαξ και ένα κράτος μέλος, για παράδειγμα, εισάγει τόνο στη χώρα. Πρέπει να κάνει κάποιες επαληθεύσεις, το τις είπα πριν. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει το έγγραφο, αν μη τι άλλο, αλλά να επαληθεύσει και το κατά πόσο είναι εντάξει το έγγραφο αυτό και κατά πόσο η αρχή που το έχει επικυρώσει είναι σωστή. Γιατί αν δεν αναφέρεται στο κατάλογο η κάτι, τότε δεν ισχύει η αρχή αυτή. Άρα δεν είναι σωστή η επικύρωση. Δεν έχει γίνει από την κατάλληλη αρχή. Είπαμε ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα προκειμένου να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες σχετικές με τις αρχές επικύρωσης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία αυτά τα μεταφέρει στην ΕΚΑΤ. Για τις τελικές διατάξεις τώρα. Όπως είπα και νωρίτερα, ο κανονισμός 4 του 2003 αναφέρεται σε διάφορα στατιστικά δεδομένα που έχουν παρακολουθήσει εισαγωγή, εξαγωγή, τριών προϊόντων. Η ΚΑΤ είχε αποφασίσει τότε να έχει τρία συστήματα για τρία διαφορετικά είδη, που είναι και ο τόνος και ο ξυφίας και ο μεγαλόφθαλμος τόνος. Τα... Για τον ξηφία δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, αλλά για τον κοινό τόνο είπαμε ότι άλλαξαν τα πράγματα από την ΚΑΤ, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να τροποποιηθεί ο κανονισμός αυτός και αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Εν κατακλείδη, σήμερα το σύστημα αυτό είναι στα πλαίσια της καταπολέμησης της παράνομης αλίας. Πέρα από τον γενικό αυτό στόχο όμως εγγράφεται και στα πλαίσια ενός νομικού συστήματος που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ξέρετε, ο κανονισμός 1005-2008 καθορίζει ένα κοινοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το σύστημα αυτό που έχει να κάνει μόνο με τον τόνο και που εγκρίθηκε από την ΙΚΑΤ, εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο του κανονισμού αυτού που καταπολεμά την παράνομη αλία εφόσον ο κανονισμός στο άρθρο 13 καθορίζει ένα σύστημα ε, προγράμματος τεκμηρίωσης ελευμάτων. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται η σύνδεση με το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλλιευμάτων που εγκρίθηκαν από ε, διάφορους οργανισμούς μεταξύ των οποίων και η ΚΑΤ. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν εγκρίνεται. Το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλλιευμάτων η ΚΑΤ θα θεωρηθεί ε, αντίστοιχο του συστήματος πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 13. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι οι διάφοροι φορείς όταν εισάγουν ή εξάγουν προϊόντα λίας δεν πρέπει να δίνουν δύο πιστοποιητικά και ε, η ΚΑΤ και η ΕΝΕΝ. Το πιστοποιητικό για το τόνο θα είναι αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπει ο κανονισμός ΕΝΕΝ. Συνεπώς, και νομίζω ότι χαίρονται γι' αυτό οι διαφοροί φορείς, θα έχουμε να διαχειριζόμαστε ένα σύστημα ενιαίο τόνου που θα συμφωνεί με τον κανονισμό μας ENN. Τέλος, χρειαζόμαστε ένα σύστημα ε, τεκμηρίωσης καινούριο, μια πρόκειται για ένα ενιαίο έγγραφο. Για τα θέματα ελέγχου πρόκειται για να ζωτική σημασία μέσο προκειμένου διάφορες αρχές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και όχι μόνο, να μπορούν να κάνουν τις επαληθεύσεις. Όλα τα συμβαλόμενα μέρη έτσι θα ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει με τον τόνο που παίρνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα, αν δεν έχετε πρόβλημα θα το δώσουμε στον κύριο Στίβενσον. τις τελευταίες ε, μέρες κάναμε πολλές συζητήσεις για τον ερυθρό τόνο και για το site της. Εγώ από ό,τι κατάλαβα στη Μεσόγειο υπάρχουν πολλές περιοχές όπου υπάρχει ερυθρός τόνος και που γίνεται αλίευση του μιλάμε για τη Μεσόγειο και μιλάμε για αλίες οι οποίοι δεν συμβιβάζονται με τους γενικούς κανόνες προφανώς ε. οπότε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κύριε Ρωμέβα, η πρώτη μου παρέμβαση πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτών που είπε ο, και ο κύριος Στίβενσον. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την παρούσα κατάσταση, αλλά αν τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει στα πλαίσια του ΣΥΤΕΣ ε, κάποια μνήα που θα αναφέρεται συγκεκριμένα στο διεθνές εμπόριο, όλα αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε ε, να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα και αυτό που είναι προφανές είναι ότι τα μέτρα τα οποία πρέπει να υιοθετηθούν, κάποια από αυτά ε, είναι εξελίξη, ε, είναι σημαντικά. Θα ήθελα να επισημάνω κάποιες πτυχές συγκεκριμένα. Καταρχάς, σε όλον αυτό τον κύκλο ε, κυρίως ε, για την πιο βιομηχανική πλευρά, αν θέλετε, της αλίευσης και της εκμετάλλευσης του τόνου, ε, μας ενδιαφέρει κυρίως το θέμα της αλίευσης. Και εδώ έχουμε μια πρώτη δυσκολία, η οποία δεν αναφέρθηκε, αλλά απαγορεύεται ρητά, για παράδειγμα, η χρήση ε, συγκεκριμένων δικτυών για να ε, επισημάνουμε πού υπάρχουν τόνοι για την αλίευσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε επιχειρήσει χρησιμοποιούν ε, τέτοια... Mm, τέτοια αεροπλάνα για να εντοπίζουν που βρίσκονται κοπάδια τόνων. Ε, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν άμεσες, μια άμεση επίπτωση σίγουρα που είναι το θέμα του ελέγχου και της εποπτείας αυτών των ε, δραστηριοτήτων θα πρέπει να εντοπίζονται και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, διότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για το φαινόμενο αυτό και υπάρχουν και αρκετέ ενημερώσεις για τα στοιχεία αυτά και θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Υπάρχει μια δεύτερη πτυχή, η οποία επίσης μου φαίνεται σημαντική. Είναι η διαφορά, το διάστημα μεταξύ ε, αλίευσης και μεταφοράς. Δεν το κάνει απαραίτητα η ίδια επιχείρηση αυτό. Το καλοκαίρι ε, ήμουνα σε παρατηρήσεις, αποστολές παρατήρησης ε, σε ανοιχτή θάλασσα. Ήμασταν στο τέλος της περίοδου της αλίευσης του τόνου και διαπίστωσα σε κάποιες περιπτώσεις πώς λειτουργούν τα πράγματα και πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες. Υπήρχε μια ομάδα η οποία αλίευε, η οποία ψαρεύει ε, εκεί στην περιοχή και αυτή τη στιγμή πλέον ο τόνος βρίσκεται στα δίχτυα, αλλάζει η επιχείρηση, αλλάζει το αλληλευτικό σκάφος και υπάρχει ένα σκάφος το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει άλλη εθνικότητα, μπορεί να έχει άλλη εντολή, μπορεί να είναι και η ίδια επιχείρηση, αυτό δεν το ξέρουμε πάντα. Ε, Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα αυτή τη συνεκτικότητα το οποίο ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει η τεκμηρίωση λοιπόν να είναι συνεκτική, να είναι συγκεκριμένη και εδώ να σα επισημάνω και κάποιον άλλον κίνδυνο τον οποίο διαπίστωσα εγώ εκεί η διεισόμαση. Μόλι ε, επικυρωθεί ένα έγγραφο, δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον σε αλλαγή του περιεχομένου του, ε, του σκάφους και σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται αυτό. Ε, πρόκειται ε, για κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου έχουμε τον τόνο που ελέγχθηκε, ο οποίος σιγά σιγά αυξάνεται μέχρι να φτάσει στον τελικό του προορισμό. Επομένως, έχουμε αυτή τη δυσκολία και δεύτερον υπάρχει και ο, η δυσκολία του ελέγχου στη θάλασσα. Όχι το, των εκφορτώσεων, αλλά των... Ε, ε, κοντέινερ που περιλαμβάνουν τον τόνο που μεταφέρεται. Θα πρέπει δηλαδή στο τέλος να γίνεται και ένας έλεγχος ε, ο οποίος θα εντοπίζει ποια είναι η διαδρομή που ακολουθήθηκε, αυτή τη στιγμή σαλιεύθηκε και πού πήγε τελικά μέχρι να φτάσει να εκφορτωθεί και αν είχαμε τη σειρά που ακολουθήθηκε. Ε, και υποθέτω ότι κανονικά με τα μέτρα που λαμβάνετε θέλετε να διορθωθεί όλη αυτή η διαδικασία, αλλά θέλουμε και το έγγραφο να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Υπάρχει και μια τρίτη πτυχή, όταν τα λεύματα βρίσκονται πλέον στα δίχτυα μπορεί να έχουμε για παράδειγμα 100 τόνους ε, τόνου σε ένα δίχτυ αλλά μπορεί να έχουμε και πάχυνση στη διαδικασία και αντί για 100 τόνους να έχουμε 150 στην τελική διαδικασία. Εδώ θέτω ερώτηση γιατί δεν το έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα δεν ε, καταλαβαίνω ποιος αποφασίζει και πώς αποφασίζουμε. Ε, είναι πολύ τεχνική ερώτηση. Πώς αποφασίζουμε λοιπόν ότι ε, ο τόνος αυτός που αλλιεύσουμε κατά 55 τόνους. Δηλαδή ε, αν αυτή η αύξηση σε τόνους είναι αποτέλεσμα πάχυνσης. Πώς το ξέρουμε. Είναι μια τεχνική ερώτηση που θέτουμε στο θέμα αυτό. Ε, ούτως ή άλλως η ερώτηση λοιπόν είναι διπλή. Πώς ε, το καθορίζουμε και ποιος είναι υπεύθυνο. Ε, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που πρέπει να το κάνει ή θα πρέπει να γίνει μια εξωτερική επιθεώρηση η οποία θα επιβεβαιώνει ότι όντως αυτή η πάχυνση ε, είναι των τόνων που αναφέρονται. Και έχω και μία ερώτηση που δεν έχει να κάνει και τόσο σχέση με τη βιομηχανική αλία, έχει να κάνει με το πιο εύκολο εντό εισαγωγικών τμήμα. Πρόκειται για τι αλλιεύσει εντός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι οι πτυχέ, αν θέλετε, οι οποίες είναι λιγότερο προβληματικές. Για παράδειγμα, έχουμε αλλιεύσει σε κάποιες περιοχές της Μεσογείου, έχουμε μικρή κλίμακα, παραδοσιακή αλληλεία ή και αθλητική αλληλεία ε, ή για ψυχαγωγικού σκοπού. Κάνοντας κάτι παράλληλο, μια παράλληλη εργασία, τον ε, κανονισμό ελέγχου, διαπίστωσα ότι υπάρχει πρόβλημα με συγκεκριμένα σημεία τα οποία καθορίζονται. Ε, αυτή είναι μια ερώτηση που προκύπτει από τον κλάδο, από μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή στη Μεσόγειο. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένας λιμένας ο οποίο έχει εντοπιστεί, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά ή αρκετά μακριά από το σημείο στο οποίο αλλιεύεται ο τόνος και ε, διευκρινίζω για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάω για βιομηχανική αλία, μιλάω για πιο παραδοσιακή αλία. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος να μην ε, πιστοποιηθεί, να μην καταγραφεί αυτή η αλία, διότι δεν ε, είναι λογικό να πάει κάποιος στο λιμένα ο οποίος έχει καθοριστεί για αυτή τη διαδικασία και ε, ουσιαστικά αυτό καταγράφεται ως ε, αλία παράνομη. Ενώ ο λιμένας ο οποίος έχει καθοριστεί ε, δεν μπορεί να κάνει την καταγραφή, θα μπορούσε ίσως να γίνεται καταγραφή σε κάποιους άλλους λιμένες ε, ανταυτού. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα έτσι. Αυτή η ερώτηση λοιπόν μου ήρθε από τον κλάδο και ήθελα να τη θέσω εδώ ως ε, ε, στα πλαίσια δηλαδή αυτής της αναθεώρησης θα ληφθεί υπόψη είναι αυτή η διαδικασία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο τώρα. Merci, ΣΥΤΕΣ και την ταξινόμηση και του ερυθρού τόνου και την πρόταση που έγινε σχετικά, αυτά δεν θα τα σχολιάσω. Το θέμα του παραρτήματος ΣΥΤΕΣ δεν είναι καινούριο. Έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια συζητήσεις ε, σχετικά και θεωρείται έχει γίνει λόγος και για απειλή εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την εμπορία και υπάρχει και το σύστημα αυτό των δηλώσεων, το πρόγραμμα αν θέλετε, δηλώσεων που έχει στόχο να ενισχύσει τους ελέγχους στην εμπορία Τώρα, δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη προβλήματα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν. Τώρα, η καταγραφή των ο, αλλιευμάτων δεν σχετίζεται με τις απειλές για την εμπορία και τα λοιπά, αλλά με την ανασύσταση του αποθέματος ε, που αποφάσισε το Συμβούλιο. Το σχέδιο, το σχετικό περιλαμβάνει όλες τις λεπτομερείς, ε, τους λεπτομερείς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και Μεταξύ αυτών των μέτρων υπάρχει και ένα σύστημα παρακολούθησης των διαφόρων φάσεων μεταφοράς του αλλιεύματος. Πρώτα, πρώτα πρώτα πρέπει να υπάρχει και το σκάφος που αλλιεύει να είναι δηλωμένο και εγκεκριμένο και η επιχειρήση το ίδιο. αν ε, δεν είναι δηλωμένες επιχειρήσεις αυτές ε, δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε σε αγορά ούτε σε πώληση τόνου προφανώς ε, και από εκεί και πέρα ε, αναφερθήκατε σε δίχτυα ή κλουβιά ή κουτιά ε, δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό ότι η επιχείρηση δεν ήταν δηλωμένη, εγκεκριμένη γιατί μου φάνηκε παράξενο τουλάχιστον αυτό που άκουσα στα γαλλικά το «κάζ» που ελέγχθη για την ε, αλληλεία του τόνου. Τώρα από εκεί και πέρα για τα αεροπλάνα, που αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τα κοπάδια του τόνου. Δείτε ε, στη Μεσόγειο φέτο και πέρσι ε, εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες ε, γίνονται έλεγχοι για τα αεροσκάφη αυτά. Το 2008 διαπιστώθηκαν παραβάσεις ε, και έγιναν σχετικές ενέργειες, οπότε κακώς χρησιμοποιούνται τα ε, αεροσκάφη αυτά, τα οποία κανονικά απαγορεύονται από τα ισχύοντα μέτρα. Τώρα, από εκεί και πέρα μεταξύ της αλλιεύσης και της α, διατήρησης αν θέλετε ή πώληση ή οτιδήποτε άλλο του, του τόνου ε, το θέμα που λέτε ε, για τη μεταφορά τι να σας πω ε, πολλές φορές μεταφορά αυτή διαρκεί εβδομάδες διότι ότι ε, πολλές φορές τα λιεύματα μπαίνουν μέσα σε συγκεκριμένα κουτιά ή τέλο πάντων κοντέινερ ε, τα οποία παραμένουν εκεί και περιμένουν ε, να έρθει κάποιος να τους ρημουλκίσει άρα πρέπει να γίνουν τόσα τον αριθμό για να τα ρημουλκίσει κάποιος περνάνε λοιπόν βδομάδες πολλές φορές και όντως μπορούν να συμβούν πολλά στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων για τη μεταφορά βεβαίως απαιτείται να αναφέρεται και ο αριθμός ε, τα στοιχεία αναγνώριση του ρημολκού σκάφους υπάρχει και η δήλωση για τη μεταφορά που και αυτή απαιτείται και γίνονται και έλεγχοι. Τι να σας πω, παρακολουθείτε και η φάση αυτή. Και οι έλεγχοι γίνονται και στη θάλασσα και στο ρημουλκό που έρχεται να μεταφέρει. Και έλεγχος των εγγράφων και έλεγχος των ε, εμπορευμάτων, ας πούμε των αλλιευμάτων. Και βεβαίω από εκεί και πέρα μπορεί ένα ρημουλκό να πάει μέχρι το σημείο Α και να έρθει ένα άλλο ρημουλκό να πάρει το ίδιο, τον ίδιο τόνο πλέον, το ίδιο αλίευμα να πάει μέχρι το σημείο Β κλπ. κλπ. Και έχουν μια σκηταλοδρομία τρόπον την αλλημουρκών. όλα αυτά παρακολουθούνται ή θα έπρεπε να παρακολουθούνται. Τώρα, τι γίνεται, ο τόνος φτάνει σε κάποιο σημείο αυτό το σημείο μπορεί να είναι σημείο ηχθειοκαλλιέργειας τρόπων την, όπου παχύνεται ο τόνος ε, άμα το έχει αλλιευθεί κάποιο ηχθής τον, την άνοιξη ε, μπορεί να παχυνθεί μέχρι το φθινόπωρο ή το τέλος χρονιάς ε, Υπάρχει λοιπόν ένα σαφέ στάδιο πάχυνσης και ο μέσος όρος πάχυνσης του ερυθρού τόνου που ε, παχύνεται σε ηχθειοκαλλιέργειες ε, είναι 26%. Τώρα μου λέτε πώς ελέγχεται η πάχυνση αυτή, τι να σας πω. Άμα φέρετε 100 τόνους τόνου σε μια εχθειοκαλλιέργεια, εγώ ξέρω μόνο τη μέση ε, τιμή πάχυνση, το μέσο ποσοστό και αν βγα... φέρετε λοιπόν 100 τόνους και πάρτε 120, εγώ θεωρώ ότι είστε μέσα στην ορμάλ πάχυνση των 26%, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, καταλαβαίνω κιόλα τι λέτε, αλλά για τον ε, για τους ελέγχους εμείς ε, εκτός από το βάρος να αναφέρεται και ο αριθμός των ψαριών είτε είναι έχουν παχυνθεί είτε όχι τα χίλια ψάρια θα παραμείνουν χίλια ψάρια Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιπλέον στοιχείο του αριθμού των ψαριών μας εξασφαλίζει και θα πρέπει οι επιθεωρητές μας να ελέγχουν και τον αριθμό των ψαριών που μπήκαν στην ηχθειοκαλλιέργεια και που βγήκαν μετά. Που μπήκαν οι απάχυνες και που βγήκαν. Τώρα, για τα συγκεκριμένα λιμάνια. Εδώ υπάρχει ένα μέτρο της ΣΥΚΑΤ, Όλα τα σκάφη ε, που αλλιεύουν ερυθρό τόνο πρέπει να τον εκφορτώνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια. Εγκεκριμένα λιμάνια. Δεν ξέρω τώρα αν ε, ε, θεωρούνται λίγα τα εγκεκριμένα μέχρι στιγμής ε, λιμάνια και μπορεί η μπορεί να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα κάτι μελη είναι αυτά που ορίζουν τα λιμάνια. Ο Ικάτ λέει ότι Ξέρουμε ότι είναι σύστημα του ΙΚΑΤ και όχι των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, μας περιορίζει και ο ΙΚΑΤ σε όλα αυτά τα πράγματα. Ορίζονται λοιπόν τα συγκεκριμένα λιμάνια από τα κράτη-μέλη. Δυστυχώ δεν υπάρχει αρκετή ευελιξία. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, κύριε Ρωμέβα, θα σας δώσω το λόγο. Ναι, ναι, για να πείτε ό,τι θέλετε, μην ανησυχείτε. Δύο επιπλέον ε, ερωτήσει έχω να κάνω. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί βλέπετε μου ήρθαν άλλε δύο ερωτήσει μετά από τι απαντήσει που άκουσα από την Επιτροπή. Η πρώτη. Υπάρχει μια πρακτική που έχει καταγγελθεί ακόμα και από τους αγοραστές στην Ιαπωνία για παράδειγμα που κατήγγειλε τη χρήση του ίδιου πιστοποιητικού για τρία διαφορετικά τμήματα, τρία διαφορετικά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι κάτι που αποτελεί την εξαίρεση, είναι ο κανόνας, γι' αυτό και σας ρωτάω. Υπάρχει δυνατότητα να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το εξαγωγικό τμήμα χρησιμοποιεί το ίδιο πιστοποιητικό. Γιατί. Μπορεί να υπάρξει διόρθωση σε αυτό. Και σας είπα, έχω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω όμως αν είναι ο κανόνας ή η εξαίρεση. Δεύτερον, ίσως να είναι και πιο προφανές, πιο συνηθισμένο, σε αυτές τις αποστολές διαπιστώνουμε πώς γίνεται η αλίευση και η μεταφορά του τόνου στη Μεσόγειο συγκεκριμένα και διαπίστωσα ότι πάντα δηλώνουν κάτω από την πραγματική αλίευση. Είναι σαν να υπάρχει άρρητη συμφωνία ανάμεσα στον αγοραστή και τον πολιτή. Υπάρχει ένα τμήμα το οποίο δεν δηλώνεται δηλαδή ρωτάω και συγγνώμη αν ακούγεται αφελής η ερώτησή μου, η ποσότητα αυτή ξέρουμε πώς είναι και υπάρχει κάποια εκτίμηση για την αξία συνολικά. Και τι μηχανισμοί υπάρχουν συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Επαναλαμβάνω, συγγνώμη για την αφελή ερώτηση, αλλά μερικές φορές βλέπετε είναι τόσο κατάφορο που πολύ καλή, πολύ καλή αφέλεια μερικές φορές κύριε Ρωμέδα. Λοιπόν, να απαντήσετε κύριε Κέμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να απαντήσω στον κύριο Ρομέδα. Πρώτα απ' όλα για τη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερε για την χρήση του ίδιου πιστοποιητικού αναφέρεται στο έγγραφο αλίευσης, ότι χρησιμοποιείται το ίδιο πιστοποιητικό για τρία διαφορετικά πράγματα. Όπως είπα και πριν, μπορεί να συμβεί, αλλά περιορισμένα. Πράγματι, μπορεί να έχετε ένα εγγραφό αλίευσης, πάντα για τους 100 τόνους που έδινα πριν παράδειγμα, που μπορεί να πάει σε κλουβί και στη συνέχεια με κομμάτια να εξαχθεί παραπέρα. Οπότε το ίδιο πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί και για τα τρία κομμάτια που θα εξαχθούν. Είναι λογικό. Και εξηγούμε στους διάφορους φορείς κάθε φορά, το λέει και ο κανονισμός, υπάρχει ένα σύστημα ενιαίου εγγράφου. Δηλαδή, αν επανεξάγεται μερικός από τους 100 τόνους, γιατί έχετε έναν Ιάπωνα πελάτη που θέλει 5 τόνους. Τι κάνετε. Παίρνετε αντίγραφο του αρχικού εγγράφου των 100 τόνων και επικυρώνετε ένα άλλο έγγραφο για 5 τόνους. Και η σύνδεση γίνεται με τον αριθμό που φέρει το έγγραφο. Δηλαδή, Έχετε το έγγραφο από την αρχική ποσότητα των 100 τόνων και της ε, ποσότητας που εξήχθη, των 5 τόνων. Προσοχή, το, η φωτοτυπή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την Εθνική Αρχή και αυτή. Δηλαδή και τους 5 τόνους πρέπει να επικυρώσετε, το έγγραφο για τους 5 τόνους, αλλά και το αντίγραφο των 100 και τα δύο. Υπάρχει δυνατότητα, προβλέπετε στο κείμενο το αντίγραφο, η φωτοτυπία και απάνω υπάρχει πάντα ο αριθμός που δείχνει ότι οι 5 ετών προέρχονται από τους 100. Τώρα για το ότι δηλώνονται λιγότερες ποσότητες, χαμηλότερες από τις πραγματικές. Είναι δύσκολο εύκολο να μιλήσουμε για μια εκτίμηση, αλλά σήμερα δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτού του είδους η πρακτική, γιατί ας υποθέσουμε ότι ένας αλλιές παίζει αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και με τη συνενοχή του αγοραστή. Τελικά, αν οι διάφοροι αυτοί οι φορείς ελεγχθούν, αλλά όχι αρκετά ώστε να έχουμε ελέγξει ακριβώς τον αριθμό των αλληλευμάτων κτλ κάποια στιγμή θα φτάσει στην Ιαπωνία η μερίδα αυτή, το κομμάτι αυτό και είναι επικίνδυνο γιατί αν έχει περάσει από όλους τους προηγούμενους ελέγχους αλλά τελικά μπλοκαριστεί στην Ιαπωνική αγορά καταλαβαίνετε ότι χάνει. Αυτός προσπάθησε να κάνει την απάτη γιατί όλοι κάνουν τους ελέγχους τους κανονικά οπότε ακόμα και αν έχει ξεφύγει από τους προηγούμενους ε, κάπου θα πιαστεί αν έχει δεκα, δεκάδες τόνους μπλοκαρισμένους στην Ιαπωνία, καταλαβαίνετε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από αυτό το διέξοδο, από αυτή την κατάσταση. Και αν δεν έχετε δηλώσει τις ποσότητές σας από την αρχή, δεν θα μπορέσετε να βγείτε από αυτό το διέξοδο. Οπότε οικονομικά δεν συμφέρει κανένα αυτό το παιχνίδι πια θα σας απογοητεύσω γιατί δεν έχουμε εκτίμηση των παράνομων ποσοτήτων αυτών. Αλλά σίγουρα καθημερινή μας δουλειά είναι να επαληθεύουμε τις ποσότητες για να δηλώνονται σωστά ελέγχοντας όλες τις πληροφορίες που παίρνουμε και από την χώρα που εισάγει το προϊόν και από τη δήλωση αλίευσης κλπ. κλπ. Με τους ελέγχους αυτούς επαληθεύουμε τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρωμέβα υποθέτω ότι ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις. Να ξαναπεράσουμε τώρα στο σημείο 9, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, που είναι η... Ε, μελλοντική ε, πολυμερή συνεργασία στον τομέα τη αλυσίας στον ε, βορειοανατολικό βορειοανατολικό ατλαντικό κυρία Καρβέλα είναι εδώ για να μας παρουσιάσει το θέμα. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πρόταση, ένα σχέδιο κανονισμού που αφορά το βορειοανατολικό Ατλαντικό. Έχει, η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο να εντάξει στο ευρωπαϊκό δίκαιο ε, ένα σύστημα μέτρων ελέγχου που εγκρίθηκε από τη ΣΕΠΑΝ, μια περιφερειακή οργάνωση αλίας. Ε, και επειδή υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις που πρέπει να τις σεβόμαστε, γι' αυτό είναι σημαντικό να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και οι δέσμευτοι κανόνων και μέτρων. Ε, έχουν γίνει ήδη αλλαγές στα μέτρα ελέγχου της ΕΠΑΝ το 2006, το 2007, το 2007 και το σχέδιο κανονισμού που προτείνουμε εν συνόψη είναι το εξής. Απ' τη μια έχουμε τις εγκρίσεις των σκαφών, έχουμε μετά τα μέτρα ελέγχου για την αλλιευτική προσπάθεια. Μετά έχουμε εποπτεία και παρακολούθηση των σκαφών για το που βρίσκονται τα σκάφη αυτά, επιθεώρηση στη θάλασσα και μετά υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τις... Ε, ε για τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρανομιών, παρατυπιών κτλ. Θέλουμε επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα στις λιμενικές αρχές να συλλέξουν κάποια στοιχεία ε, τα οποία ε, ελιμενίζονται, τα στοιχεία για τα σκάφη που ελιμενίζονται εκεί και για τη σημαία υπό την οποία κινούνται. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο για την ε, για να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη παράνομη αλία υπάρχει εκεί στα πλαίσια αυτής της αλίας μια διάταξη παρόμοια με αυτή που σας λέω τώρα όπου το, οι λιμενικές αρχές μπορούν να ζητούν στοιχεία για την σημαία που έχει το πλοίο το σκάφος. Αυτά κυρία Πρόεδρε με δύο λόγια για το σχέδιο κανονισμού που ελπίζουμε να εγκριθεί ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ε, pues no Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, αυτή η έκθεση θεωρητικά έχει δοθεί στην πρόεδρο επειδή δεν το ήθελε καμία πολιτική ομάδα. Ε, ξέρω ότι απλά μεταφέρουμε στην κοινοτική νομοθεσία μία απόφαση που έχει ληφθεί αλλού. Επομένως θα το μελετήσουμε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρβέλα. Και... Με αυτό νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα διάφορα. Σημείο 15. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι από τα διάφορα. Σημείο 16. Δεν σας είδα. Κύριε Ριμπελίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα διάφορα, επειδή αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση της νέας ε, θητείας της ε, του Κοινοβουλίου. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που συναντιόμαστε για να οργανώσουμε τις εργασίες μας. Διαπίστωσα ότι στους ε, παλιούς φακέλους, ε, στην παλιά θητεία, προσέχουν ιδιαίτερα το θέμα της ε, διατήρησης των δινδών, ε, των συστημάτων αλληλείας ε, και της μέρημνας για το περιβάλλον. Διαπιστώνω εδώ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να κάνω και λάθος γιατί είμαι νεοεκλεγής. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την υγεία των καταναλωτών, των Ευρωπαίων δηλαδή που καταναλώνουν αυτά τα ψάρια και πολύ συχνά στις, ε, στα τραπέζια της ε, Ευρώπης δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Διακόπτη, Πρόεδρος. Θα ήθελα να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν ξέρουν από πού προέρχονται αυτά τα ψάρια που τρώνε. Τι τρώνε. Και αν αυτό το ψάρι είναι από μολυσμένες ε, θάλασσες, η Μεσόγειος αλλά και άλλες ε, θάλασσες ε, αυτή τη στιγμή βιώνουν ε, κάποιες στιγμές αν θέλετε δυστυχείς. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν στην Επιτροπή μας στον προγραμματισμό των επομένων ετών να λάβουμε υπόψη και το θέμα αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να καθορίσουμε με κάποιο τρόπο την προέλευση όλων αυτών που βρίσκουν οι, πολίτε, ε, οι πολίτες στα τραπέζια τους. Ακριβώς για την μέρημνα της υγείας τους. Ε, κατανοώ ότι αυτό μπορεί να είναι κοινή αρμοδιότητα με άλλες επιτροπές, αλλά πιστεύω ότι η Επιτροπή Αλίας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιολογήσει και να δει αυτό το θέμα. Κατανοώ επίσης, ε, διότι εγώ είμαι από μια πολιτική εμπειρία της Ιταλίας που είναι τελείως διαφορετικά τα κοινοβουλευτικά θέματα. Καταλαβαίνω ε, πώς είναι δυνατόν η ακραία γραφειοκρατία με κάποιο τρόπο να διευκολύνει αλλά και να δυσχεραίνει το έργο της, ε, ε, των κοινοβουλευτικών εργασιών. Θα πρέπει όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να βρουν και μια λύση, να περάσουμε λίγο πέρα από αυτή την ε, κρύα και σκληρή γραφειοκρατία. Θα πρέπει εμείς ως Ευρωβουλευτές να το υπερκεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Η ερώτησή σας είναι πολύ ευστοχή και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Η υγεία δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αυτό όσον αφορά στι αρμοδιότητε. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που όντω είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτροπή μα και είναι το θέμα τη ετικετοθεσίας. Η ετικετοθεσία προβλέπεται από την κοινή οργάνωση αγοράς, ε, ε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε κανονισμούς, ε, σαφώς θα μπορούσαμε να τον βελτιώσουμε τον κανονισμό, αλλά υπάρχουν κανονισμοί και αυτό το οποίο αποτελεί πρόβλημα είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν τηρούν την κοινοτική νομοθεσία για την ετικετοθεσία. Υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με αυτό που αναφέρατε εσείς και είναι το θέμα της οικολογικής ετικέτας. Εγώ ήμουν και εισηγήτρια και είχαμε είχαμε κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας για, την, ε, για τις οικολογικές ετικέτες για να μπορέσουμε να προσπίσουμε και τους καταναλωτές. Ε, προς έκπληξή μας, στο τέλος της προηγούμενης θητείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νομοθετική πρόταση για τις οικολογικές ετικέτες οριζόντιου χαρακτήρα που κάλυπτε όλα τα θέματα της ε, οικολογικής ετικετοθεσίας και πέρασε στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εγώ τότε ήμουν συντονίστρια του ΕΛΚ και πολέμησα για αυτό το θέμα, πραγματικά ε, έγινε έξω φρενών, διότι ήταν ένα θέμα το οποίο αφορούσε τον τομέα της αλίας, έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, διότι η βιωσιμότητα της αλίας δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα άλλων τομέων, για παράδειγμα με τα υποδήματα ή με οτιδήποτε άλλο, και θεωρούσαμε ότι αυτό το θέμα δεν έπρεπε να περάσει έτσι. Το θέμα πέρασε στη συναπόφαση και τελικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία, γιατί εγώ δεν δεχόμουν σε καμία, με καμία κυβέρνηση να γίνει το θέμα αυτό ε, οριζόντιου χαρακτήρα. Ε, νομίζω ο κύριος Σταβάρα, ένας σοσιαλιστής ήταν αυτός ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό από πλευράς Επιτροπής Περιβάλλοντος, κατάλαβε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα για την Επιτροπή Αλίας και καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό ε, ο οποίο ήταν ο εξή. Αφήσαμε να περάσει η δεύτερη ανάγνωση, αλλά υπήρχε ρητή γραπτή δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεσμεύθηκε να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη πρόταση για την αλληλεία, η οποία θα ήταν ε, αρμοδιότητα τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνσης που ασχολείται με θέματα αλληλεία. Πριν από το τέλο του έτου, υπάρχει ένα κατάλογο θεμάτων με τα ε, οποία θα συζητήσω με τον κύριο Φωτιάδη. θα συζητηθούν αυτά και στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται και αυτό το θέμα και το τι αποφασίστηκε τότε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω αν ήμουν αρκετά σαφή στην εξήγησή μου, αλλά σε σχέση με αυτό που σας είπα, σας εξήγησα πώς εργαζόμαστε. Φυσικά, κάθε φορά που θα υπάρχει αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, ε, θα δούμε τι γίνεται. Μπορεί να υπάρχουν ίσως και κάποιες εκθέσεις πρωτοβουλίας που είναι πιο δύσκολες, αλλά το θέμα της ετικέτας είναι κάτι το οποίο είναι έτοιμο και είναι μία από τις δυνατότητες που θα μας δοθούν να συζητήσουμε και αυτό το θέμα που σας απασχολεί. Υπάρχει κοινοτική νομοθεσία για, την, ε, για τις ετικέτες και σας λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει κανονισμός, είναι ότι δεν τηρούνται από τα κράτη-μέλη τα όσα καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. Και φυσικά είναι ανησυχητικό το θέμα, διότι οι καταναλωτές αγνοούν τι ψάρια τρώνε. Εγώ είμαι νοικοκυρά, πηγαίνω στο ψαρά και βλέπω ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες νοικοκυρές. Έχω μια κάποια πείρα, ε, ξέρω ότι ε, μπορεί να λέει ότι έχουμε καλαμάρι από μια περιοχή και είναι από οποιαδήποτε άλλη περιοχή παρά ε, από την περιοχή που λέει ότι είναι. Υπάρχει και το Παγκάσιος που έρχεται από συγκεκριμένη περιοχή. Ε, για μένα είναι πολύ σοβαρό το θέμα αλλά οι περισσότερε νοικοκυρέ το αγοράζουν, το θεωρούν πάρα πολύ νόστιμο, δεν έχει αγκάδια και το τρώνε τα παιδάκια. Ε, και εμεί δεν ξέρουμε ούτε που το ψαρέψαμε, ούτε που το βρήκαμε αυτό το παγκάσιο. Τα παιδάκια όμω το τρώνε, δεν έχει αγκάδια και επομένω στην Ισπανία θεωρείται το καλύτερο ψάρι τι προσπαθώ να σας πω, ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί και εγώ θα σας υποστηρίξω. Αλλά η επόμενη μας μάχη είναι όντως το θέμα της οικολογικής ετικοτοθεσίας και οποιαδήποτε πρωτοβουλία από πλευράς ομάδος σας, που είναι και δική μου, θα μελετηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κύριος Στίβενσον. Αυτά που μόλις τώρα είπατε κυρία Πρόεδρε, που σχετίζονται και με τον καυγά που είχαμε τελικά με την Επιτροπή Περιβάλλοντος μου θυμίζουν και κάτι τι άλλο. Η Επιτροπή Ανάπτυξης όπως ξέρετε ε, έχει ε, λόγο σε σχέση με τη Συμφωνία ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Γουινέα. Θα γνωμοδοτήσει λοιπόν παρόλο που εμείς είμαστε αρμο... αρμόδιοι η αρμόδια επιτροπή. Ε, εμείς θέλουμε να συζητηθούν και να μελετηθούν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης γενικότερα. Σύμφωνα, αυτός είναι ένας καυκάς που κάναμε πάντα και εγώ ήμουνα ε, τότε και εισηγήτρια για ένα θέμα για την ε, Δυτική Αφρική και είχαμε και ένα μεγάλο καυγά με την Επιτροπή Ανάπτυξης, θα το θυμάστε και αυτό όσοι ήσασταν εδώ. Το θέμα για την Επιτροπή ανάπτυξη είναι πολύ σαφέ. Η Επιτροπή ανάπτυξη θέλει να ασχοληθεί με ένα θέμα που δεν την αφορά και ε, δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε γνωμοδοτήσεις εσείς, τα, οι προθεσμίες είναι λίγο δύσκολες, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε εταιρικέ ε, συμφωνίες αλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αλίας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει πολλά πράγματα να κάνει άλλα, τα οποία δεν τα κοιτάνε καθόλου και ασχολούνται με τα δικά μας. Έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος εδώ που συμμετέχει και στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Εγώ ε, έχω μπει και αναπληρώτρια στην Επιτροπή Ανάπτυξης και να ασχοληθώ και με αυτά τα θέματα. Δεν θα επισέλθω τώρα σε όλες αυτές τις ιστορίες, δεν είναι τις παρούσεις. Ε, μου είπε και ο γιατρός να μην αγχώνομαι. Ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ παρόλα αυτά θα πάω στην Επιτροπή Ανάπτυξης. δεν ξέρω, ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δεν ξέρω τι είναι, ε, θα πάω να τον βρω, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση, να συνεργαστούμε, να εργαστούμε θετικά και να προσπαθήσουμε να μην ε, μπαίνει ο ένας στα χωρικά είδατα του άλλου. Υπήρχε και μια πρόταση της κυρίας Λεβάν να δούμε και τι γίνεται με τα θέματα της Επιτροπής Ανάπτυξης που ασχολείται με θέματα που είναι δικά μας. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα θέματα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να λυθούν με την πρόταση που κάνουμε για την επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων. Κύριε Ρεμπελίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Διότι και αυτό το μαχητικό σας πνεύμα, κυρία Πρόεδρε, μου δίνει πραγματικά την αίσθηση ότι η γραφειοκρατία που πολλές φορές ε, δυσκολεύει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω ο γιατρός να σας δώσει το πράσινο φως, να μπορέσετε να παλέψετε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και πιστεύω ότι μία μάχη για να διαφυλάξουμε τους πολίτες, διότι διαπιστώνω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνεται μια ιδιαίτερη προσοχή για να σώσουμε τα πάντα εκτός από τους πολίτες. Όλα τα είδη των ζώων, το περιβάλλον, τα φυτά, και ουσιαστικά τους πολίτες τους ξεχνάμε. Πρέπει όμως να ξεκινήσουμε από τους πολίτες. Αυτό το μαχητικό πνεύμα μου δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι στη διάθεσή σας για το δικό μου γιατρός μου λέει ότι πρέπει να τσακώνομαι συχνά με όλους για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου λέει όχι, αλλά μην νομίζω ότι θα κάνω μόνο ότι μου λένε οι γιατροί. Έτσι κι στην οικογένειά μου είχα πάντα γιατρού, ποτέ δεν του έδινα σημασία. Τέλο πάντων, τώρα προσπαθώ να του ακούω, αλλά θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Ωραία, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, επόμενο σημείο που είναι οι ανακοινώσει σχετικά με τι αποφάσει που λήφθησαν χθε του συντονιστέ. Ε, αποφασίσαμε για την κυρία Λεβέν στους συντονιστές, ε, κάτι που εκείνη ζήτησε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα σας τα στείλω για να τα ξέρετε. Και έτσι περνάμε στο 17ο και τελευταίο σημείο στη Μέση που είναι η ημερομηνία τη επόμενη συνεδρίασης που θα είναι στι Βρυξέλλες 30 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Α, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ναι, εγώ να σας πω ότι στο έγγραφο το οποίο μας παραδώσατε, δεν ξέρω μέσω ποιας ψηφοφορία έγινε αυτή η διαδικασία και δεν ξέρω και πώς συζητήσατε το θέμα. Αποφασίσατε όμως να αποκλείετε τους αντιπροέδρους από τις συνεδριάσεις των συντονιστών. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται εν ίδια ανακοίνωσης ε, ως επικύρωση. Εγώ θα ήθελα να ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια, να περιλαμβάνουν και τους άλλους αντιπροέδρους ε, επιτροπών, διότι αυτή είναι η μία απόφαση, η μόνη απόφαση της Επιτροπής. Σήμερα το πρωί ε, είδα τι γίνεται στις άλλες επιτροπές. Στις υπόλοιπες επιτροπές οι αντιπρόεδρες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ε, συντονιστών. Αλλιώς, τι δουλειά έχουν οι αντιπρόεδροι. Διότι αν πρέπει να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο, θα πρέπει να το κάνουν και να είναι ενημερωμένοι. Αν είναι αντιπρόεδρο απλά για να κάθονται εδώ, στο έδρανο ψηλά, δεν υπάρχει λόγος, ε, αδειάζουμε και τη γωνιά και πάμε παραπέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι η διαχείριση και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της Επιτροπής μας θα πρέπει να τα μοιραζόμαστε περισσότερο. Η κατευθύνσεις της Επιτροπής θα πρέπει να είναι συλλογικές, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες Επιτροπές. Επομένως, εγώ σας ζητώ να μην επικυρώσετε την απόφαση ε, να γίνει και μια πρώτα συζήτηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να ξανασυζητηθεί η απόφαση αυτή και να δούμε τι γίνεται συνήθως. Ε, δεν ξέρω αν οι άλλοι αντιπρόεδροι θέλουν να είναι ευγενεί και να ακούσουν την ε, απόφασή σας. Εγώ θα ήθελα να γίνει μία μάχη για το θέμα αυτό, διότι σε όλες τις άλλες επιτροπές αυτό ισχύει. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιο να πάρει τη θέση μου όμως, γιατί εγώ δεν θα ήθελα απλώς να είμαι εδώ και να κάνω το πιόνι. Εντάξει, μπορούμε να μην εγκρίνουμε αυτή την απόφαση, να περιμένουμε. Καλύτερα να μιλήσετε με τις ομάδες σας, γιατί τι να σα πω. Εγώ χτε δεν ψήφισα και θέλω να το ξέρετε αυτό. Ε? Ο καθένα ε, ψήφισε, οι πολιτικέ ομάδε θα σα εξηγήσουν γιατί ψήφισαν όπω ψήφισαν. Στον κανονισμό προβλέπεται η συνεδρία των συντονιστών και προβλέπεται η δυνατότητα ή όχι να δεχτούμε του αντιπρόεδρους. Οπότε εγώ δεν φταίω, είναι απόφαση που πήραν χτε οι συντονιστέ. Εγώ σας είπα ότι θα το θέσω το ζήτημα αυτό γιατί σας το υποσχέθηκα. Και όντω το έθεσα. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήτανε. Δεν θέλω να σας πω τώρα ακριβώς τι ήταν η συζήτηση, πάντως ρωτήστε τις πολιτικές σας ομάδες γιατί ψήφισαν όπως ε, ψήφισαν. Μην το λέτε σε μένα. Όχι, μια στιγμή, μια στιγμή, γιατί είναι και ο κύριος άλλος αντιπρόεδρος εδώ που θέλει το λόγο. Οπότε, να τα βρείτε με την πολιτική σας ομάδα. Εδώ υπάρχει μία μόνο συντονίστρια. Τι να σας πω. Α, ναι, ναι, α, ναι, δεν τον είδα. Ναι, ναι, σωστά. Δεν είναι όμως οι υπόλοιποι συντονιστές εδώ. Οπότε, πρώτα να μιλήσετε με τις πολιτικές σας ομάδες και αφού μιλήσετε μαζί τους, θα δείτε. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω από πριν. Τι, δεν έχετε εμπιστοσύνη να σας εκπροσωπήσω. Εν πάση σίγουρα αυτό που δεν μπορώ να πω είναι ότι δεν πήραμε την απόφαση που πήραμε χθε. Την πήραμε. Με συνένεση, μιλήστε λοιπόν με την πολιτική σα ομάδα και θα δούμε. Να πάρουμε όσο γίνεται καλύτερη απόφαση. Συμφωνώ. Τι να σας πω, εγώ σα μεταφέρω τι αποφάσεις τι οποίες καταλήξαν χθε οι συντονιστέ. τίποτα άλλο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν αφισβητούμε καθόλου το γεγονός ότι εσείς δεν ευθύνεστε για την απόφαση αυτή. Προς Θεού. Αλλά επειδή θέλουμε η Επιτροπή αυτή να αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία, νομίζω ότι δεδομένων των όσων συμβαίνουν, η Επιτροπή Γεωργίας που κινδυνεύει να πάρει ένα κομμάτι της αλίας, εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την Επιτροπή αυτή αλίας, συμφωνούμε όλοι με αυτό. Και να τη διευρύνουμε όσο γίνεται στα θέματα που αφορούν τη θάλασσα το γεγονός ότι οι αντιπρόεδροι να μπορούν να συμμετέχουν στη διάσταση των συντονιστών είναι κάτι το οποίο βέβαια με συνένεση πρέπει να αποφασίσουμε. Αλλά εγώ συμφωνώ, τι να σας πω. Συμμερίζομαι τις απόψεις των ε, συναδέρφων. Συμφωνώ μαζί τους, ε, κύριε Στίβενσον. Πρόεδρος, δεν θέλω εδώ πέρα να τραβήξει η συζήτηση αυτή για πολύ. προφανώς και έχετε άλλη άποψη εσείς, αλλά εγώ δεν θέλω να πιέσω κανέναν, ούτε δεν θέλω να τσακωθεί κανένας με κανέναν. Προσπαθώ να λύσω τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, μιλήστε πρώτα με την πολιτική σας ομάδα και πάρτε μια απόφαση, οπότε στην επόμενη συνεδρίαση συντονιστών οι συντονιστές να ξέρουν τι να προτείνουν. Να έχουν την άποψη που έχουν και οι αντιπρόεδροι εδώ. Συγγνώμη, εγώ μιλάω τώρα, ε. σας έδωσα το λόγο, τώρα μιλάω εγώ. Μη με διακόπτετε. Λοιπόν, Νομίζω ότι αυτό πρέπει πρώτα να κάνετε, να μιλήσετε με την πολιτική σας ομάδα. Μιλήστε με τους συντονιστές σας. Επιχειρηματολογήστε. Οπότε στην επόμενη συνεδρίαση συντονιστών θα μεταφέρουν ό,τι έχουν να μεταφέρουν. Εγώ θα συνεργαστώ με τους συντονιστές και θέλουν να υπάρχει συνένεση. Ορίστε κύριε Μιλάνα, σας ακούω τώρα. Εγώ σας βλέπω πολύ νευρική κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ πολύ ήρεμα το θέτω το θέμα. Δεν ξέρω αν εχθές, γιατί δεν ήμουν παρόν, οι συντονιστές ψήφισαν αυτή τη θέση. Στα πρακτικά δεν προκύπτει. Μου λένε ότι συμφώνησαν με τη θέση της Προέδρου. Εσείς δεν ψηφίσατε, αλλά προτείνατε να μην συμμετέχουν οι αντιπρόεδροι στη συνεδριά των συντονιστών. Αυτό είναι το θέμα. Ε, καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να ε, ε ξαναπεράσετε το θέμα στις πολιτικές ομάδες. Από πλευρά μου, εγώ θα κάνω ακριβώ αυτό που προτείνετε εσεί. Αλλά θα ήθελα να σα ζητήσω πριν από την προηγούμενη συνεδρίαση να μην επικυρώσετε αυτή την ψηφοφορία. Οι υπόλοιπε αποφάσει μια χαρά είναι κατά την άποψή μου. Δεν... Θα ήθελα να μην επικυρώσετε αυτό το σημείο και να το αναβάλλετε για μια επόμενη συζήτηση. Ε, με πολύ ηρεμία, χωρίς κανέναν εκνευρισμό, διότι πραγματικά εγώ θεωρώ ότι κάνω κάτι χρήσιμο για τις εργασίες της Επιτροπής, όπως ελπίζω ότι το ίδιο θεωρούν και οι άλλοι αντιπρόεδροι και ε, οι συμμετέχονται στην Επιτροπή. Αλλιώς ε, δεν κάνουμε τίποτα. Καθορίζουμε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, αλλά δεν μπορεί να διαφέρει από Επιτροπή σε Επιτροπή, διότι αφού είμαστε όλοι ευρωβουλευτές, εγώ το θέτω θέμα ισορροπίες. Ούτε πρωταγωνιστής θέλω να γίνω, ούτε να πάρω τα ημία από κάποιον άλλον. Αλλά θέλω να συνεργαστούμε, ε, με πάθος και με αποφασιστικότητα. Αυτό και μόνον αυτόν. Κύριε Στίβενσον. Δεν θέλω να γίνει μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα, αλλά στο παρελθόν πάντα έτσι κάναμε μόνο συντονιστές και όχι αντιπρόεδροι. Οι αντιπρόεδροι εμφανεί σε έκτακτες περιπτώσεις όπου υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλο θέμα, τότε αποφάσισε το Προεδρείο της Επιτροπής. Πάντως ανέκαθεν οι συντονιστές συνεδρίαζαν. Γιατί διορίζεται κάποιος συντονιστής για ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να καθίσει να κάνει αυτή τη δουλειά που γίνεται με την κατανομή της εργασίας κλπ. Αν τώρα από εκεί και πέρα ε, θέλουμε ε, να διευρύνουμε την ομάδα, να έχουμε όλους τους συντονιστές από τις διάφορες ομάδες, να έχουμε και όλους τους αντιπρόεδρους και τα λοιπά. Είναι σαν να συνεδριάζει η Επιτροπή ολόκληρη ξανά. Μέχρι τώρα δηλαδή οι συναντήσεις των συντονιστών ήταν της τάξης των 30 λεπτών. Άμα ε, είναι πολύ άριθμη η συνάντηση τότε θα πάρει και πολύ περισσότερο χρόνο. Δύο λόγια θέλω να σας πω. Τις αποφάσεις που πήραμε χτες σας τις είπα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ψηφίσαμε. Με απόλυτη πλειοψηφία. Δεν θέλω να σας πω ποιος ήταν υπέρ και ποιος κατά από τους συντονιστές, αλλά γι' αυτό σας λέω μιλήστε με τους συντονιστές σας οι οποίοι θα σας εξηγήσουν τι και πώς. Εγώ εδώ δεν θα αποκαλύψω τίποτα, με απόλυτη πλειοψηφία πάντως. Έτσι, για τους λόγους που εξήγησε και ο κύριος Στίβενσον και άλλοι. Μιλήστε λοιπόν με τους συντονιστές σας, άμα θέλετε το αφήνουμε σε κρεμότητα αυτό το θέμα αλλά δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό για όλο. Λοιπόν, μιλήστε με του συντονιστέ σα και στην επόμενη συνεδρίαση θα δούμε αν έχει αλλάξει η άποψη. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εγώ δεν την πήρα αυτή την απόφαση. Οι συντονιστέ την πήρανε. Μου ζητήσατε να το θέσω, το έθεσα. Θα μπορούσα και να μην το θέσω, γιατί ποτέ δεν είχαμε στους συντονιστές και τους ε, αντιπρόεδρους. Ξέρω ότι άλλες επιτροπές κάνουν αλλιώς. Αυτό το θέμα λοιπόν παραμένει σε κρεμότητα και στην επόμενη συνεδρία, αφού έχετε μιλήσει με τους συντονιστές σας, θα προχωρήσουμε. Σας λέω, σας ανακοινώνω τις αποφάσεις που πήραν οι συντονιστές χτες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Οι υπόλοιπε εγκρίνονται όμως οι αποφάσεις οι υπόλοιπες. Ε? Ευχαριστώ, για σας.